I think we can start. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich eröffne die Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Είναι η τελευταία συνεδρίαση μετά τις καλοκαιρινές ε, διακοπές. Ελπίζω να περάσετε καλά και να επανέλθετε καλύτερα. Έχουμε κάποιους ε, φιλοξενούμενους από την κάτω Σαξτονία. Είναι 70 μέλη από, από την περιοχή αυτή ε, που έχουν έρθει σήμερα να παρακολουθήσουν εδώ. Και επίσης έχουμε και έναν άλλο ε, πολύ καλό καλεσμένο. Είναι η εκπρόσωπος ε, των πρασίνων της, του κρατηδίου αυτού, η Ζουζάνε Μέγκε. Καλώς ήρθατε. Η ημερήσια διάταξη λοιπόν ε, εγκρίνεται αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Από ό,τι βλέπω δεν υπάρχουν και αν δεν υπάρχουν μπορούμε να εγκρίνουμε και τα πρακτικά της 5ης Ιουνίου του 2016. Δεν έχω κάποια ανακοίνωση ως πρόεδρος. Πάμε τώρα στην πρώτη ανάγνωση για τις τεχνικές προδιαγραφές ε, για την ε, εσωτερική ναυσιπλοεία. Η Βομπέλετ είναι η Ιβο Μπέλετ είναι εισηγητής. Εδώ πρόκειται για τις τεχνικές προδιαγραφές εσωτερικής ναυσιπλοείας και πρέπει σύμφωνα με τον κανονισμό να ξεκινήσει η συνάντηση σήμερα μιλώντας για τη διαδικασία. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου στις 22 Ιουνίου στην Ολομέλεια ε, κατέστησε γνωστή την ανακοίνωση του Συμβουλίου για τις προδιαγραφές αυτές σύμφωνα με το άρθρο 66 παράγραφος 2 του κανονισμού ε, πρέπει η θέση του Συμβουλίου να τεθεί ως πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνάντησης και συνεδρίασης της, ε, της ε, Αρμόδιας Επιτροπής ε, που ακολουθεί αυτήν την ανακοίνωση. Έτσι λοιπόν σήμερα στην Επιτροπή μας, επειδή έχει κατατεθεί αυτή ε, κατατέθηκε αυτή η θέση του Συμβουλίου και ξεκινάμε αυτό, η δεύτερη ανάγνωση. Ο εισηγητής ε, σήμερα το απόγευμα θα μας ε, δώσει κάποια στοιχεία για αυτή τη δεύτερη ανάγνωση. Έχουμε 1η Σεπτεμβρίου την ψηφοφορία. Εδώ ήταν για ενημέρωσή σας αυτό το σημείο. Τώρα έχουμε Μαριάν Μαρινέσκου ως εισηγητή για το επόμενο σημείο, το σημείο 5. Πρόκειται για τις ε, τροπολογίες, ε, για τον ε, πρόταση κανονισμού ΕΑΣΑ της Κομισιόν το Μάη. Ο εισηγητής, ο κύριος Μαρινέσκου, μας παρουσίασε τις 861 επιπλέον προτάσεις τροπολογίας των συναδέλφων και του δίνουμε τώρα το λόγο για να μας εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη. Κύριε Μαρινέσκου. Ευχαριστώ πολύ. Όντως πρόκειται για 861 τροπολογίες, οι 100 περίπου ήταν δικές μου. Είμαι ευγνώμων γιατί περίμενα πάνω από 2.000. Φτάσαμε περίπου στις 1.000, άρα είμαι ικανοποιημένος. Ε, έχω εξετάσει αυτές τις τροπολογίες λίγο πολύ, όχι με μεγάλη λεπτομέρεια, λίγο πολύ, νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε σχεδόν παντού συμβιβαστικές λύσεις. Κάποιες, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ καλές ιδέες. Νομίζω λοιπόν ότι μαζί μπορούμε να φτιάξουμε μια πολύ καλή έκθεση. Εγώ θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις μόνο για κάποια λίγο αντιφατικά ζητήματα της υπηρεσίας εδάφους, το ground handling και της ε, την εξοπλισμό των αεροδρομίων που είναι κρίσιμο για την ασφάλεια. Είναι κάποιες ε, τροπολογίες οι οποίες θέλουν να βγει τελείως η πιστοποίηση. Να πω ότι ε, ο σύνδεσμος των εταιριών που ασχολούνται με τις υπηρεσίε εδάφους υποστηρίζουν αυτή την πρόταση, διότι μιλάμε απλώς για μία δήλωση από έναν οργανισμό. Ελπίζω λοιπόν ότι θα φτάσουμε σε ένα συμβιβασμό που θα είναι υπέρ της βιομηχανίας. Μπορώ να, του κλάδου δηλαδή. Ελπίζω να σας πω ότι ακόμα και το αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης υποστηρίζει αυτή την πρόταση για να καταλάβετε. Εξεπλάγει βέβαια διότι υπάρχουν και πολλές ε, τροπολογίες που ε, ε, αντικαθιστούν τις πράξεις κατά με εφαρμοστικές πράξεις. Εμείς στο Κοινοβούλιο πάντοτε υποστηρίζαμε τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση, γιατί έτσι μπορούμε να δώσουμε τη γνώμη μας, αλλά ελπίζω ότι θα δείξουμε κατανόηση. Επίσης, για την πιστοποίηση του προσωπικού που ασχολείται με τα ηλεκτρονικά της αναέρειας κυκλοφορίας, η ΕΑΖΑ έχει ήδη κάποια έγγραφα με αυτή την πρόταση. Υπάρχει επίσης μια άλλη αντίφαση η εθελούσια μεταφορά ευθυνών Κάποιοι ζητούν πιο σκληρή λύση, άλλοι θέλουν να είμαστε πιο χαλαροί. Υπάρχουν και κάποιες τροπολογίες που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια. Είναι η εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας του ΕΑΖΑ μάλλον στην ασφάλεια. Πάντοτε θα μπορούσαμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Ε, εγώ, αν θέλετε τη γνώμη μου, ένα διοικητικό όργανο θα ήθελα, ε, εκτελεστικό συμβούλιο, ε, με μικρό αριθμό ανθρώπων, όχι 28 ας πούμε άτομα. Αυτή είναι η πρότασή μου για τα τέλη μεταφορά μέρους των τελών από την Γεροκοντρόλ στον ΕΑΖΑ. Να πω ότι το 2009 η ρυθμιστική δραστηριότητα για την, ε, για την ενέργεια κυκλοφορία πέρασε από το Eurocontrol στην ΕΑΖΑ και τώρα ε, θέλουμε να κάνουμε και το ίδιο και με αυτή την περίπτωση. Αυτό ήταν που είχα να πω. Να πω, λέει ο Πρόεδρος, ότι σήμερα δεν έχουμε χρόνο. Αύριο θα συζητήσουμε αυτό το θέμα πιο αναλυτικά. Οι σκιώδεις έχουν δύο λεπτά και ένα οι υπόλοιποι. Καμπριέλε Πρόης είναι εκτός ο μιλήτρια. Έχουμε σημειώσει αρκετή πρόοδο κατά του τελευταίου μήνε και πολλέ από τι τροπολογίε που κατατέθηκαν ε, καταδεικνύουν ακριβώ ότι πολλοί συνάδελφοι έχουν ασχοληθεί επισταμμένω με αυτό το ζήτημα. Θα ήθελα εκ των να σας ευχαριστήσω για την πολύ καλή συνεργασία που θα έχουμε και είχαμε ήδη. κάποια ζητήματα κεντρικής ε, σημασίας έχουν ήδη τεθεί στο πλαίσιο τροπολογιών από συναδέλφους από άλλες πολιτικές ομάδες ε, και ήδη σε κάποια σημεία υπάρχει, υπάρχουν ενδείξεις ε, ε, συνένεσης μεταξύ των διαφόρων πολιτικών ομάδων και σας ευχαριστώ όλους για αυτό το ε, γεγονός. Ε, ως εγώ ε, επιχαίρω το γεγονός ότι ε, πολλοί από εμά ε, ε, ασχολούμαστε με το ζήτημα των κοινωνικών πτυχών. Ε, όπως σας έχω πει επανειλημμένα αυτό το ζήτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μένα προσωπικά και για την πολιτική μου ομάδα και θεωρώ ε, πως είναι απαραίτητο να βελτιώσουμε ουσιαστικά την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, δηλαδή αυτές οι συμβάσεις ε, περιορισμένη διάρκειας θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να βελτιωθούν. Ε, σε ό,τι αφορά τις επίγες, την επίγεια κυκλοφορία, ε, και τι σχετικές υπηρεσίες. Βλέπω ότι υπάρχουν διστάμενε απόψει μεταξύ των ε, πολιτικών ομάδων. Ε, Εμεί θεωρούμε πως θα πρέπει να προβούμε σε κάποιε αλλαγέ. Όπω φαίνεται και από τι δικέ μου τροπολογίε, Για παράδειγμα, το προσωπικό για τη διασφάλιση, που είναι αρμόδιο για την ασφάλεια στου αερολιμένου, θα πρέπει να καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογή αυτού του κανονισμού. Θα ήθελα να ζητήσω από του υπόλοιπου συναδέλφου να υποστηρίξουν αυτέ τι προτάσει Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το τομέα Τη της ασφάλειας ε, στις αερομεταφορές ε, βλέπω ε, πως πολλοί συνάδελφοι θεωρούν πως θα πρέπει να αναλάβει έναν κάποιον σημαντικό ρόλο η ΆΣΑ αλλά από την άλλη πλευρά εγώ παραμένω σκεπτική εάν θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την δυνατότητα η ΕΑΣΑ να μπορεί να δίνει δεσμευτικού χαρακτήρα κατευθυντήριες γραμμές. Επίσης δεν γνωρίζουμε ή αμφιβάλλουμε κατά πόσο θα μπορούσε να επεκταθεί η εντολή, η σχετική εντολή της ΕΑΣ. Οπότε ε, θα ήθελα να ε, υποστηρίξω την τροπολογία ε, της συναδελφού Λουσεβά για την τροπολογία 67. Επίσης θα πω ότι είμαι υπέρ τη διαγραφή του σημείου F σιγματάφ, δηλαδή από το άρθρο 109, παρότι γνωρίζω ότι κάποιοι συνάδελφοι έχουν αντίθετη άποψη. Κατά τελευταία μα συνεδρίαση, η Επιτροπή μα είχε ανακοινώσει ότι θα προβεί σε μια ακριβή περιγραφή και διαφοροποίηση ε, των αρμοδιοτήτων τη Eurocontrol ε, και τη ΕΑΣΑ. Ε, μια τέτοια αναλυτική περιγραφή θα μα βοηθούσε πολύ ούτω ώστε να μπορέσουμε να βρούμε να φτάσουμε στου κατάλληλου συμβιβασμού. Για μα είναι πολύ σημαντικό να φτάσουμε σε μια συνένεση η οποία θα μπορέσει να λάβει υπόψη και τα συμφέροντα των μικρότερων ε, φορέων ε, και ενδιαφερομένων ε, στον τομέα τη αεροπορία. Σε ό,τι αφορά τα μοντέλα αεροσκαφών, αυτά θα πρέπει να δείχνουν διαφορετική μεταχείριση από τα μη επανδρομένα, από τα drones. Δηλαδή και κάτι ακόμα σε ό,τι αφορά τη διατύπωση, να πω ότι θεωρώ πως ο νέος κανονισμός είναι τόσο σημαντικός ε, ούτως ώστε να μην ε, είναι απαραίτητη ή ενδεδειγμένη, εν πάση περιπτώσει, η ενδεδειγμενη λέξεων όπως κατάλληλο, ελάχιστο, ενδεδειγμένο και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Πέντε ποντά. Έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από τη δική μας πλευρά θα ήθελα να πω πως οι τροπολογίες ε, που ανέφερε μόλις ε, τώρα η κυρία ε, Πρόησε σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τις συμβάσεις περιορισμένου χρόνου εργασίας να πούμε ότι πραγματικά αποτελεί ένα σκάνδαλο το τι συμβαίνει αυτή την περίοδο στον τομέα της αεροπορίας και νομίζω πως η ε, σχετική τροπολογία ε, ε, τη κυρία Επρό κινείται προ σωστή κατεύθυνση και θα ήθελα να την υποστηρίξω εξ ονόματο τη πολιτική μου ομάδα. Εγώ υπέβαλα κάποιε τροπολογίε από τη δική μου πλευρά, ειδικότερα σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο 5 και την διαγραφή του από τον κανονισμό που προτείνει η πρόταση. Δηλαδή, έτσι όπω προβλέπεται εκεί η ίδρυση του σχετικού οργανισμού είναι λανθασμένη. Ναι, προφανώς μπορούμε να κάνουμε κάποιες βελτιώσεις στο υφιστάμενο πλαίσιο, αλλά το να προτείνουμε να δημιουργήσουμε μια ε, εκτεμελίων νέα υπηρεσία, ένα νέο οργανισμό είναι κάτι το λαθασμένο και θα ήθελα να το εξετάσουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι ω ενδεχόμενο να διαγράψουμε δηλαδή αυτή την πρόταση. Από εκεί και μετά άλλε πτυχέ είναι πολύ θετικέ, δηλαδή υπάρχει μια εποπτεία, μια παρακολούθηση από την πλευρά των αρμόδιων εθνικών αρχών ε, ε, και από την πλευρά τη οπότε αυτά ε, στο πλαίσιο του συστήματο πραγματικά είναι επαρκή. Ευχαριστώ, λέει η Ευχαριστώ. Ε, δεν υπολόγιζα ότι θα πάρουμε τόσο γρήγορα το λόγο γιατί υπάρχουν και δεν, νόμιζα ότι δεν υπήρχαν νόμιζα ότι υπήρχαν περισσότερες σκιώδεις εισηγητές. Α, ναι, Ματίας έχει το ε, λόγο σκιώδης εισηγητές, ε, το συγγνώμη που τον ξέχασα επειδή συνήθως κάθεται δίπλα σας, ε, γι' αυτό δεν τον είδα. Ναι, η βιομηχανία ο κλάδος δηλαδή της αεροπορίας χρειάζεται ένα πλαίσιο το οποίο να είναι και συμμετοχικό και ε, σταθερό και νομίζω ε, πως ε, και αυτό εκφράζεται και στην πρόταση που κάνει η ίδια η Επιτροπή σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση του Οργανισμού Ασφάλειας για την Αεροπορία. Άρα λοιπόν εγώ θα ήθελα να επιμείνουμε στην διατύπωση της πρότασης της Επιτροπής και να περιοριστούμε σε ό,τι αφορά τις τοπολογίες που θα καταθέσουμε. Ας εστιάσουμε λοιπόν στα κύρια ζητήματα και βέβαια γι' αυτό με ε, ε, εκπλήσει το γεγονός ότι ο συνολικό αριθμό είναι 1103 τελικά τροπολογίε οι οποίε κατατέθηκαν. Ε, νομίζω πω ε, δεν θα πρέπει εδώ να ασχοληθούμε με ζητήματα όπω ο βάρο των μη επανδρομένων ε, οχημάτων αέρα, των drones δηλαδή, αλλά πιο σημαντικά ζητήματα είναι ε, το πεδίο εφαρμογή που θα καλύπτει η ΆΣΑ, ποια είναι η ασφάλεια που θα διασφαλίζει και ούτω καθεξή. Άρα λοιπόν νομίζω πω η ασφάλεια, ο προπολογισμό και η ασφάλεια σε ό,τι αφορά και τα drones είναι τα τρία σημαντικά που θα πρέπει να μα απασχολήσουν. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, νομίζω πω η ΑΣΑ θα πρέπει να έχει το δικαίωμα τη πρωτοβουλία σε ό,τι αφορά τα ζητήματα ασφάλεια, ειδικότερα κυβερνοασφάλεια, αλλά ε, και των ε, ζητημάτων ε, διέλευσης αεροσκαφών πάνω από ζώνες σειράξεων. Άρα λοιπόν θεωρώ πως θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα το δικαίωμα να δει δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές σε ό,τι αφορά τη διέλευση από ζώνες σύραξης ειδικότερα μετά από το σχετικό τραγικό δυστύχημα που είχαμε και νομίζω πως θα πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με αυτό το ζήτημα δηλαδή ε, τη ε, διέλευση αεροσκαφών από τέτοιε ζώνε σύρευση και θα ήθελα να καλέσω του συναδέλφου ε, από τι υπόλοιπε πολιτικέ ομάδε να υποστηρίξουν αυτέ τι τροπολογίε για να μην έχουμε, μία, να έχουμε ένα ενιαίο μέτωπο έναντι του Συμβουλίου. Μετά, σε ό,τι αφορά τι μοιρασμένες αρμοδιότητες. Ε, νομίζω πως θα πρέπει ε, να είμαστε πολύ σαφεί εδώ σε ό,τι αφορά την κατανομή των αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο του προπολογισμού και νομίζω πως ο δικός μας κανονισμός θα πρέπει να είναι βασικός ε, και να λειτουργήσει ω μια εργαλειοθήκη, δηλαδή να μας δίνει μια σειρά από, από διαφορετικά εργαλεία τα, οποία θα μπορεί να αξιοποιεί η ΕΑΣΑ. Και σαφώ θα πρέπει να υπάρχει καθαρός, σαφής διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ Eurocontrol ε, και EASA και ακριβώ η EASA να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ω toolbox. Από εκεί και μετά σε ό,τι αφορά τα drones, ναι, χρειαζόμαστε ασφάλεια και ταυτόχρονα και ευελιξία βέβαια, γιατί υπάρχουν ε, και ταχύτατες εξελίξει στον τομέα της τεχνολογίας ε, και επειδή έχουμε ακριβώ εδώ νομοθετικέ πράξει που είναι κάτω εξουσιοδότηση, θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στις λεπτομέρειες. Δηλαδή, ο εισηγητής έχει τη δυνατότητα να οργανώσει μια μικρή εκδήλωση τεχνικού χαρακτήρα γιατί υπάρχει και ένα πρωτότυπο ήδη το οποίο ε, έχει δημιουργηθεί σε ό,τι αφορά αυτές τις κατεξουσδιώτες πράξεις και με βάση το οποίο μπορεί να ε, διατυπωθεί και σχετική πρόταση για την ΕΑΣΑ και έχουμε ζητήσει και από τον κύριο Μαρινέσκου ε, να μας ενημερώσει ως προς το πώς ακριβώς το μελλοντικό δηλαδή κανονιστικό πλαίσιο θα λειτουργήσει στην πράξη. puheenjohtaja. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον εισηγητή για την πολύ καλή πρόταση έκθεσης. Όπου ήδη ακούσαμε αρκετά σε σχέση με την αρχική πρόταση. Έχουμε καταθέσει μια τροπολογία που θα θέλαμε να συζητήσουμε μαζί σε σχέση με την αεροπλοεία. Γιατί είναι σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη μας την ασφάλεια όσον αφορά την εργασία, γιατί σχετίζεται άμεσα με τις συνθήκε εργασίας αυτό. Οπότε οι συνθήκες εργασίας είναι ένα ζήτημα το οποίο μας ε, αφορά και το οποίο διασφαλίζει την ασφάλεια στην αεροπλογία. Γι' αυτό θα πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη μας και γι' αυτό το λόγο έχουμε καταθέσει κάποιες προτάσεις. Έχουμε θεσπίσει την ιδέα του pay to fly που μπορεί κανείς να αποδεχτεί ή όχι. Σημαντικό λοιπόν θέμα η ασφάλεια, αλλά νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγουμε τις περιπλοκές, τις υπερβολικά μεγάλες και δύσκολες για τους επιβάτες. Επίσης θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την έρευνα και την ανάπτυξη, ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις διαδικασίες ασφάλειας. Έχουμε επίσης και μία τροπολογία που αφορά όλους τους εμπλεκόμενους στον κλάδο αυτό και που τους επιτρέπει για τους εργαζόμενους πριν ξεκινήσουν τη δουλειά τους να γίνονται κάποιοι έλεγχοι όσον αφορά θέματα ασφάλειας ώστε αυτό να έχει επιπτώσει και στην ασφάλεια των επιβατών για το executive boarding αυτό δεν το πολύ κατάλαβα ομολογώ θα ήθελα κάποιος να μου το εξηγήσει για να δούμε τι γίνεται. Εμείς δεν θέλουμε πάντως να υπάρχει γραφειοκρατία. Αυτό πρέπει να αποφευθεί οπωσδήποτε. Εξάλλου, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να αλλάξουν εδώ και πολλά πράγματα σε σχέση με αυτό που κάνουμε μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρίως που τηρήσατε το χρόνο. Είναι πολλοί που θέλουν να μιλήσουν, όμως ο χρόνος είναι μόνο ένα λεπτό για τον καθένα. Ο κύριος Κόχ. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Μαρινέσκου για την εξαιρετική πρόταση. Έχω καταθέσει πολλές τροπολογίες, οι τρεις έχουν να κάνουν με το γερμανικό κείμενο, το οποίο έχει πάρα πολλά ε, λάθη. Ε, ε υπέρ της ε, ανάπτυξης της ΕΑΖΑ και της αντιμετώπισης ε, των ε, προκλήσεων πρέπει να αποφύγουμε αλληλοεπικαλύψεις. Για το ground handling πρέπει να δρά η ΕΑΣΑ, αλλά να ασχολείται μόνο με την ασφάλεια και δεύτερον να πρέπει, θα πρέπει να βοηθά στην τήρηση των διεθνών προδιαγραφών για αυτό το θέμα είναι σημαντικό να έχουμε ξεκάθαρη νομοθεσία. Αν θέλει ούτως ή άλλως η Κομισιόν να βάλει το θέμα των ε, μοντέλων, ε, να βγάλει μάλλον το θέμα των μοντέλων ε, και να μπει στο κανονισμό, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το θέμα επίσης αυτό που με απασχολεί ιδιαίτερα είναι αυτά τα πτυτικά μέσα που χρησιμοποιούνται για τη διάσωση. Νομίζω ότι έχει ήδη δοθεί πάρα πολύ μεγάλη αρμοδιότητα. Υπάρχουν και ιδιώτες που εκπληρώνουν αυτές τις υπηρεσίες και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Το τελευταίο σημείο έχει να κάνει με το παράρτημα το οποίο έχει να κάνει με την ηλεκτρονική κίνηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Τσιγητή και τους Κιώδης και θα ήθελα να υπογραμμίσω τα εξή. Καταρχάς είναι σημαντικό να ασχοληθούμε με το θέμα της ασυλίας των, του προσωπικού της Υπηρεσία, όπως αντίστοιχα συμβαίνει και με τη συνδρομική αρχή. Θα πρέπει λοιπόν στον κανονισμό να υπάρχει μια διαδικασία που αφορά την άρση της ε, ασυλίας στα πλαίσια του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης θεωρώ ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ένα άρθρο το οποίο θα επιφέρει την υποχρέωση που θα ακολουθεί τις σωστές πρακτικές που θα απορρέουμε από την εθνική νομοθεσία. Επίσης για τις ε, εθνικές αρχές θα πρέπει οτιδήποτε αλλάζει να ενημερώνεται το προσωπικό και επίσης για τις περιβαλλοντικές περιγραφές αυτές θα πρέπει να τηρούνται απαρέκλητα και για την κοινωνική διάσταση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει βεβαίως την διαβούλευση αλλά και, την, και τον περιορισμό των έμεσων μορφών εργασίας που μειώνουν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ που τηρήσατε το χρόνο, κύριε κυρία Γκεζίνα Μάιζερ. Επιτέλους θα η ώρα μου. Ευχαριστώ. Ήθελα να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις, κάποια πράγματα που ήδη έχουν υποθεί και θα ήθελα να υπογραμμίσω. Φέτος ε, Υπάρχει αυτός ο κανονισμός, η ρύθμιση και βλέπουμε πώς θα θεσπιστεί και πώς θα έχει δυνατότητα δράση στο μέλλον η, ε, ο ΕΑΖΑ. Και γι' αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία που πρέπει να τηρούνται. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τη μεταφορά των ε, αρμοδιοτήτων για την ασφάλεια, για τα drones, ε, για τους ε, ιδιώτες, διότι πρέπει εμπορικά να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν και ατυχήματα. Και όλο αυτό είναι σωστό, όμως υπάρχουν και πολλές άλλες αρμοδιότητες που πρέπει να πάνε σε αυτή την υπηρεσία. Και θεωρώ ότι ε, έχοντας την Eurocontrol από τη μία και την, τον ΕΑΖΑ από την άλλη, καλό θα ήταν να διασφαλίσουμε την ε, συνεργασία. Ας μην έχουμε μια υπεραρχία όπως έχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει καλή συνεργασία. Ευχαριστώ. Καρίμα Ντέλη. Ένα λεπτό. Πρόεδρε, θα είναι δύσκολο να πω αυτά που θέλω σε ένα λεπτό. Πάντως, με την πρώτη ανάγνωση Νομίζω θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τη μέθοδο εργασία μας. Να δούμε δηλαδή κατά πόσο θα πρέπει να υπάρξουν ομάδες εργασίας που θα εξετάσουν τις επιπτώσει των πτήσεων των drone για να αποφύγουμε τις πολεμικέ. Να σας πω πάντως ότι η ομάδα μου βεβαίω ασχολήθηκε με τα περιβαλλοντικά θέματα, είχαμε την COP21, εξετάσαμε αυτά τα ζητήματα, είπαμε ότι η αεροπλοεία βεβαίω είναι ο πρώτο καταναλωτή ορυκτών καυσίμων, υπεύθυνο για μεγάλο ποσοστό ρήπων. Συζητάμε λοιπόν για την έσα και εξετάζουμε φιλόδοξα και αισιόδοξα σενάρια όσον αφορά το τομέα της αεροπλοείας και τη μείωση των εκπομπών. Και λέμε επίση ότι τέλος πάντων θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα για να υλοποιηθούν όλα αυτά. Να πω όμω ότι έχουμε και το κοινωνικό ζήτημα όπου εντάξει θα βρούμε κάποιες συμβαστικές λύσεις αλλά να προκαταβάλω ότι η υπαπασχόληση είναι ένα ζήτημα το οποίο επιβαρύνει την ασφάλεια γιατί έχουμε συνθήκες εργασίας υπερβολικά επιβαρημένες πιλότων και άλλου λοιπού προσωπικού. Έχουμε πιλότους με ελάχιστη κατάρτιση οι οποίοι νοικιάζονται όλες, Όλα αυτά λοιπόν έχουν επιπτώσεις σε διάφορες υπηρεσίες όπως η εξυπηρέτηση εδάφους και σε άλλες υπηρεσίες. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ώστε να πετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και νομίζω ότι σύντομα θα επανέλθουμε σε αυτά τα ζητήματα. Πιστεύω πάντως ότι για τα drone θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με το νέο σύστημα πιστοποίησης των συσκευών που συνοδεύονται από κάποιο πιστοποιητικό απόδοση και εκεί θα πρέπει να δούμε ακριβώ πρόεδρε λοιπόν λεπτομέρειε τι πρέπει να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ η Μαρία Κριστίνα Νοτού τώρα. Ευχαριστώ. Συμμερίζομαι πρόεδρε την άποψη του αδέλφου Βαντάλεν που λέει ότι πράγματι σε αυτές τις τροπολογίες τις εκατοντάδες τα ζητήματα ουσίας δεν θίγονται και νομίζω ότι οι αρμοδιότητες της ΕΑΣΑ μας κάνουν να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να υπάρχει μια αποτελεσματική και σωστή λειτουργία αυτής της υπηρεσίας, αποφεύγοντας επικαλύψεις με άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες και κυρίως θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την διασφάλιση της αρετής αυτής της ευρωπαϊκής, της επικουρικότητας. Νομίζω ότι αυτή η υπηρεσία θα έχει αρμοδιότητες, αλλά δεν θα πρέπει να γίνει αυτό ει βάρος των υπολείπων χώρων μελών. Ευχαριστώ. Ο Μιχαλ Καλά, für Flugsicherheit. Ευχαριστώ ε, και εμείς ε, υποστηρίζουμε αυτή την ε, προετοιμασία, την προσπάθεια προετοιμασία του κλάδου τη Αεροπορία για τι αλλαγέ που θα προκύψουν στα επόμενα χρόνια και βέβαια εν ώψη και τη αυξανόμενη εναέρη κυκλοφορία. Ωστόσο, εγώ υιοθετώ κριτική άποψη ω προ τι προτάσει που γίνονται για τη διεύρυνση τη εντολή και των αρμοδιοτήτων τη ΕΑΣΑ, πέραν δηλαδή αμυγός των ζητημάτων ασφαλεία. για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το περιβάλλον ε, και τον τομέα της security. Ε, δεν θεωρώ δηλαδή ε, πως η ΕΑΣΑ θα πρέπει να αναλάβει αρμοδιότητες οι οποίες ήδη ανήκουν σε άλλους και σε σχέση με τις οποίες ήδη έχουμε επιτύχει καλά αποτελέσματα. Γιατί για παράδειγμα να αναλάβει αρμοδιότητες στον τομέα των υπηρεσιών, των επίκαιων ε, υπηρεσιών υποστήριξη, ποια προστιθέμενη αξία θα έχουμε. Από εκεί και μετά, σε ό,τι αφορά τι ε, επιπρόσθετε ε, διατάξει ασφαλεία, σε ό,τι αφορά τον εξόπλισμο για τα aerodromes, θεωρώ πω μέχρι στιγμή δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα ασφαλεία. Και νομίζω πως το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο στο, της δηλαδή της, Διεθνούς υπηρεσίες πολιτική Αεροπορίας είναι επαρκές. Από εκεί και μετά τα συστήματα διαχείρισης της ε, αεροπορίας ε, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι είναι ε, συμβατά. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε κάτι παραπάνω. Δηλαδή τα υφιστάμενα συστήματα ε, ε, είναι ήδη προσαρμοσμένα στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα, οπότε μια ε, πιστοποίηση δεν είναι απαραίτητη εδώ. Δεν θεωρούμε πως η επίλυση τέτοιων προβλημάτων θα πρέπει να αποτελέσει αρμοδιότητα της ΕΑΣΑ και δεν θεωρώ πως θα πρέπει να λάβει κάποιο μέρος των κοντιλίων του Ιερου Η Λούση Άντερσον, λέει τώρα πρόεδρος, έχει το λόγο υπάρχει ένας ε, λόγος εδώ βάσιμος για τον οποίο υπάρχουν πάνω από χίλιες ε, ε, τροπολογίες. Και ποιος είναι αυτός, ότι είναι μια, ένα, πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό κανονισμό καθώς θα θέσει πρότυπα σε όλο αυτό τον κλάδο τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και πέραν αυτής. Οπότε πραγματικά είναι απαραίτητο να γίνει μια τέτοια συζήτηση και θα πρέπει να επιτύχουμε την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των κατεξοδότηση πράξεων και των εκτελεστικών πράξεων. Γιατί αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να μην επισέλθουμε σε πάρα πολύ τεχνικά ζητήματα, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν πολλά τεχνικά ζητήματα τα οποία έχουν πολιτική χρειά. Και υποστηρίζουμε τα όσα υπόθηκαν ε, από κάποιου ε, συναδέλφου, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την ε, βιωσιμότητα αυτών των μέτρων από πλευρά περιβάλλοντο. Αλλά θα ήθελα να ευστήσω την προσοχή σα σε ένα σημείο. Θα ήθελα να εξετάσει την ε, τροπολογία 363 ε, που αφορά ε, τα ζητήματα μοδιότητας των ίδιων των επιβατών, το οποίο αφορά και κάποια σχόλια που έγιναν από την Πάτη Κοινού και άλλους. Δηλαδή, θα πρέπει ο κανονισμός να υποστηρίζει την ανάληψη των σχετικών ευθυνών από πλευρά των επιβάτων σε ό,τι αφορά τον, την ασφάλεια και ταυτόχρονα διασφαλίζει την κατάλληλη νομοθεσία για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Άρα λοιπόν, η εμπιστοσύνη των επιβατών στο σύστημα είναι κέρια σημασία. Ευχαριστώ λίγο Ο Μάρκο Πίπα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Υπάρχουν πολλά καλά στοιχεία στην έκθεση. Καταρχάς να θυμίσω ε, στους συναδέλφους που διαμαρτύρονται ε, για τις τροπολογίες να πω ότι είναι πάρα πολλές από τις τροπολογίες που έχουν να κάνουν με τη διπλή αρμοδιότητα και την αλληλοεπικάλυψη γιατί δεν πρέπει ο ΕΑΖΑ να κάνει διπλή δουλειά. Να πω ε, για την πιστοποίηση, θα πω λέξεις κλειδιά. Είναι η πιστοποίηση ένα θέμα το οποίο ε, θα, πρε... θα γίνει καλά σε κάποιους ε, τομείς γιατί υπάρχουν κανόνες. Χρειαζόμαστε δεν χρειαζόμαστε αρμοδιότητες στη ΖΕΑΤΖΑ στις έκτακτες περιπτώσεις ε, ή στην ασφάλεια των πτήσεων. να πω ότι για τα τέλη ήδη και για το ground handling υπάρχουν ζητήματα κοινωνικά που φύγονται. να μην μπει ο ΕΑΖΑ, πρέπει να προσέξουμε όμως σε αυτά που ήδη υφίστανται ως κανονισμό. Επίσης για τα μεγάλα αεροδρόμια και τα μικρά αεροδρόμια πρέπει να υπάρχει κάποια ρύθμιση ώστε να μην έχουμε γραφειοκρατία που ε, να, να μην διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία τους. Κυρία Γιάλα, ευχαριστώ πρόεδρε. Εύχομαι καλή επιτυχία στον εισηγητή, ο οποίο είναι εργασιομανή για τι τροπολογίε. Υπάρχει μια τάση εξευρωπαϊσμού του κλάδου. Και αυτό για τις μεταφορές στα πλαίσια των ομαδιοτήτων νομίζω ότι αυτές θα πρέπει να γίνουν στην ΕΑΣΑ. Επίσης, για τη συνεργασία με το Eurocontrol και αυτή είναι σημαντική. Όπως επίσης και η ανάγκη, εκτός από το περιβάλλον και την ασφάλεια, επειδή σχετίζεται άμεσα με την ασφάλεια, να λάβουμε υπόψη μας σοβαρά τα κοινωνικά ζητήματα. Θυμάστε το ατύχημα της German Wings και άλλες περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με κοινωνικά ζητήματα υγεία των τοποργασία. Επίσης, το προσωπικό. Καμπίνας. Και αυτόν τα δικαιώματα θα πρέπει να προστατεύονται. Όπως επίσης και τον εργαζομένων στο κάργο. Έχουμε ένα κλάδο ο οποίο αυξάνεται συνεχώς. Αυξάνεται και η ευθύνη του, οπότε θα πρέπει να συνεχίσουμε τον διάλογο στο να αποφύγουμε δυσάρεστες εκπλήξεις και αποτελέσματα. Για τη φορολογία τώρα. Νομίζω θα έχουμε μία έκθεση από την Επιτροπή Λόγου του Προβλησμού, πάνω στην οποία θα πρέπει να δουλέψουμε και εμείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τώρα η Τζάκη Φώστερ ένα λεπτό όμως, γιατί μετά έχει δύο λεπτά ο εισηγητής. Ευχαριστώ. Να ζητήσω συγγνώμη από τον εισηγητή. Είχα καθυστέρηση δύο ώρες με την πτήση μου από το Μάντσεστερ. Κάτι που δεν σχεδίαζα φυσικά, γιατί αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό για μένα. Δεν είχα καμία πρόθεση να δω 1100 τροπολογίες. Έχω φυσικά καταθέσει πολλές από αυτές, διότι έλαβα υπόψη πολλά σχόλια σχετικά με τις υπηρεσίες ενέργειας κυκλοφορίας από τους κατασκευαστές, ε, τις αεροπορικές εταιρείες και άλλα. Δεν ήμουν εδώ για να ακούσω τα αρχικά σχόλια του κυρίου Μαρινέσκου, όμως είπαμε κάποια πράγματα στη συνάντηση των σκιωδών σχετικά με την ονομασία του οργανισμού. Να την αλλάξουμε δηλαδή. Και υπήρξε και ένα στοιχείο που είχε να κάνει με το funding και το cross-funding από το Eurocontrol. Νομίζω λοιπόν ότι για προφανείς λόγους ε, δεν έπρεπε να, δεν μπορούμε να αλλάξουμε, όπως και το cross-funding. Επίσης, για, την, για το ground handling πρέπει να παραμείνουν τα στάνταρ που ήδη λειτουργούν καλά. Έχω καταθέσει 75 τροπολογίες και ελπίζω ο εισηγητής, επειδή υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, και επειδή πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν πρόκειται για ένα έγγραφο κοινωνικής πολιτικής, αλλά για ένα έγγραφο ρυθμιστικό, κανονιστικό που πρέπει να προσαρμοστεί στις επιταγές των καιρών και επειδή θέλουμε ένα αποτελεσματικό έγγραφο, ελπίζω ο εισηγητής να λάβει υπόψη κάποια από τα σοβαρά σχόλια που έκαναν οι και άλλοι. Θα βοηθούσε πάρα πολύ και έτσι ελπίζω ότι θα φτάσουμε και σε κάποιο συμπέρασμα. Και εμείς στο ECR περιμένουμε, με αδει... αδειμονούμε για τις ε, συμβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ. Γιάννης Νίλσον, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ ειδικότερα στο ζήτημα της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων άλλων οργανισμών στον ΕΑΣΑ. Αυτό σημαίνει ότι ε, δηλαδή οι εν λόγω εργασίες ήδη εκτελούνταν από αυτές τις ε, ε, υπηρεσίες ή τους οργανισμούς και με αυτή την μεταβίβαση τι κάνουμε ουσιαστικά μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες οι οποίες ήδη εκτελούνταν αποτελεσματικά από αυτούς τους οργανισμούς. Από εκεί και μετά θα πρέπει να ξέρουμε ότι επειδή ακριβώς πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό τομέα θα χρειαζόμαστε μια ισχυρή εντολή και έχουμε από τη μία πλευρά μια αρμόδια αρχή για τον εθνικό αναέριο χώρο στα κράτη-μέλη και από την άλλη πλευρά έχουμε την ΕΑΣΑ ως συναρμόδια αρχή. Ε, αλλά βέβαια όταν υπάρχουν δύο τέτοιοι φορεί που είναι και οι δύο αρμόδιοι, υπάρχει δυσκολία στο να ληφθεί μια κοινή απόφαση. Όταν δηλαδή λαμβάνει μια απόφαση η εθνική αρμόδια αρχή, δεν θα μπορεί να παρισφρέει η ΕΑΣΑ, έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν σε σχέση με αυτό το ζήτημα θα πρέπει να έχουμε μια πολύ κατηγορηματική διατύπωση. Ευχαριστώ, ε, λέω ο Πρόεδρος. Ε, θα δώσω το λόγο και στην Επιτροπή. Αλλά να πω κάτι στη συζήτηση πάτε, λέμε αυτά είναι τεχνικέ λεπτομέρειε μα λέτε ε, και ότι γι' αυτό θα κάνουμε μια κατεξουδότηση πράξη. Εμεί στο Κοινοβούλιο αποφασίζουμε κατά πόσο πρόκειται για τεχνικό ή πολιτικό ζήτημα. Γιατί αυτό είναι και το δικαίωμα μα με, με βάση τη συνθήκη τη Λισαβόνα όπω έγινε και με την έκθεση Μπένετ. Ε, ε, αγωνιστήκαμε για καιρό αλλά τα καταφέραμε τελικά. Οπότε θα ήθελα πραγματικά ε, προκειμένου να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μα α είμαστε πολύ αυστηροί. Γνωρίζουμε δηλαδή ποια πρακτική ακολουθούμε και η Επιτροπή και το Συμβούλιο προσπαθούν δηλαδή να μας περιθωριοποιήσουν στο πλαίσιο αυτών των διαδικασιών. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα πρέπει να τους αφήσουμε να το κάνουν αυτό. Θα πρέπει εμείς να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε το δικαίωμα που έχουμε να αποφασίζουμε τι αποτελεί τεχνικό ζήτημα και τι αποτελεί πολιτικό ζήτημα και βέβαια η Επιτροπή μπορεί να σχολιάσει αυτά τα ε, τεχνικά ζητήματα που πλευρά τη συμπαρέμβαση που θα κάνει τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τον κύριο Μαρινέσκου και για το γεγονό ότι μα δίνετε το λόγο σε ό,τι αφορά ε, το πού βρισκόμαστε σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Καταρχήν ε, χαιρόμαστε για το γεγονό ότι πραγματικά επιτυγχάνουμε ταχεία πρόοδο σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα ε, και παρότι υπάρχει ένα, ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός τροπολογιών, η γενικότερη αίσθηση είναι ότι υπάρχει ευρεία υποστήριξη προς αυτή την πρόταση της Επιτροπής και ελπίζουμε ε, πως μέσα στις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες θα ε, καταλήξουν σε κάποιες ε, συμβαστικέ τροπολογίε, όλε αυτέ οι πολλέ τροπολογίε, οι οποίε θα είναι και πολύ χρήσιμε για την βελτίωση του κειμένου. τώρα, χωρί να θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειε, θα έχουμε ούτω ή άλλω τη δυνατότητα να επισέλθουμε σε αυτέ σε μεταγενέστερο στάδιο και για να πούμε με ποιε συμφωνούμε και ποιε όχι, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια επιμέρου στοιχεία. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντο, α μην ξεχνάμε ότι ήδη αυτό το ζήτημα συγκαταλέγεται στι αρμοδιότητε τη ΕΑΣΑ. Δεν αλλάζουμε δηλαδή πολλά σε αυτό το τομέα. Αυτό που προσπαθούμε να αλλάξουμε είναι ότι, ναι, επί τη αρχή ακολουθούμε όλου του περιβαλλοντικού κανόνε τη ΕΚΑΟ, αλλά από εκεί και μετά θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να ε, έχουμε διατάξει να ρυθμίζουμε ζητήματα περιβαλλοντικού χαρακτήρα πέραν αυτών που ρυθμίζει η, η, ΚΑΟ και βέβαια να υπάρχει και δυνατότητα παρέκκληση από αυτού του κανόνε όπω ισχύει ούτω ή άλλω και σε όλου του άλλου κλάδου αεροπορία στον κόσμο. Από εκεί και μετά σε ό,τι αφορά το, την κοινωνική διάσταση. Αντιλαμβανόμαστε ποιο είναι το σκεπτικό, η συλλογιστική αυτών των τροπολογιών, ε, αντιλαμβανόμαστε τι ανησυχίε των ε, εκπροσώπων των ε, οσοδιών των πληρωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από εκεί και μετά βέβαια είναι περιορισμένα τα όσα μπορούν να γίνουν εδώ. Ε, δεν υπάρχει δηλαδή νομική βάση που να μας επιτρέψει να ε, επιστρέψουμε σε, σε τομείς εργασιακού δικαίου ή κοινωνική ασφάλισης αλλά από εκεί και μετά κατά τη διατύπωση διατάξεων ασφαλείας ναι, ασχολούμαστε με ζητήματα όπως η κοινωνικη ασφαλεια αλλα απο εκει και του πληρώματος, η υγεία του πληρώματος, το μέλλον του πληρώματος οπότε αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει και στο πλαίσιο του νέου κανονισμού. Μετά σε ό,τι αφορά τα ντρόν, θα μία οχήματα ε, που αποτελούν και μία από τις βασικές καινοτομίες αυτών ε, τον νέο κανονισμό. Εμείς υποστηρίζουμε λοιπόν και ενισχύουμε την φιλοσοφία που έχουμε θετήσει μέχρι τώρα, δηλαδή να αναπτύξουμε μία ισχυρή αγορά για ντρόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν υποστηρίζουμε κατά συνέπεια τροπολογίε οι οποίε εξαιρούν ορισμένα τμήματα αυτή τη αγορά από το πεδίο εφαρμογή ή αλλάζουν και επαναφέρουν ουσιαστικά τον, ε, το κείμενο του κανονισμού στην κατάσταση που ισχύει σε εθνικό επίπεδο. Δεν είναι αυτό ο στόχο μα. Αντιλαμβάνομαι προφανώ ότι υπάρχουν κάποια ερωτήματα από την πλευρά του Κοινοβουλίου. Ε, ρωτάτε δηλαδή ποιοι είναι οι κανόνε που θα ισχύσουν εδώ. Δεν θέλετε να υπάρχει ένα υπερβολικά συστατικό κανονιστικό πλαίσιο. Και πράγματι, ναι, θα υπάρξει ένα ε, πρωτότυπο κανονισμό ο οποίο ε, θα διατυπωθεί από την ΕΑΣΑ και θα δημοσιευθεί στο εγγύ μέλλον, ώστε να έχετε όλοι σα μια εντύπωση ω προ το πώ θα λειτουργήσουν τα πράγματα και έτσι ε, ελπίζουμε βέβαια ότι θα συμβαστούν οι ανησυχίε σα. Από εκεί και μετά εκφράστηκαν και κάποιε απόψει σε ό,τι αφορά τι σχέσει ε, με τη Eurocontrol. Όπω είπε ο κύριο Μαρινέσκου, δεν ε, προσδίδουμε νέε αρμοδιότητε σε άσα στον τομέα του ελέγχου. Αυτό το κάναμε στο 2009. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε τώρα αντιθέτω είναι η δυνατότητα χρηματοδότηση κάποιων από αυτέ τι δράσει μέσω αυτών των τελών. Αλλά αυτές, αυτά τα τέλη δεν ανήκουν στην Eurocontrol, ε, ανήκουν σε όλους οι οποίοι ε, συμμετέχουν σε αυτό το τομέα τη ρύθμιση κυκλοφορίας, δηλαδή και, και στις αρχές των κρατών μελών και ούτω καθεξής. Ε, άρα λοιπόν, ο στόχος εδώ είναι να συνεχίσουμε τη να υπάρχει δυνατότητα της εφαρμογής του user base. Ε, της αρχής user base. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις διαφορετικές ε, ε, αρμοδιότητες, εδώ το ζητούμενο είναι να ορίσουμε τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα της ΕΑΣΑ και όχι της Eurocontrol. Άρα, κατά συνέπεια, οποιασδήποτε τροπολογίες κατευθούν σε σχέση με ρύθμιση των αρμοδιοτήτων της Eurocontrol θα είναι προβληματικές. Από εκεί και μετά σε ό,τι αφορά το σαφή διαχωρισμό μεταξύ αρμοδιοτήτων ΕΑΣΑ και Eurocontrol έχουμε ένα συγκεκριμένο roadmap, ένα οδικό χάρτη δηλαδή πορείας, ο οποίος θα δημοσιευτεί μέσα στο φθινόπωρο και ο οποίο ελπίζουμε να, να σα δώσει την απαραίτητη σαφήνεια ω προ αυτό το διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ ΕΑΣΑ και Eurocontrol. Ε, και βέβαια, εάν υπάρξουν ακόμα εκρεμή ζητήματα, μεταξύ, σε ό,τι αφορά τι αρμοδιότητε μεταξύ ASA και Eurocontrol, αυτό θα πρέπει να γίνει μεταξύ ακριβώ σε συνεννόηση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Eurocontrol απευθεία. Σε ό,τι αφορά τώρα το προπολογισμό, επιχαίρουμε την ε, ευρεία υποστήριξη που υπάρχει ω προ την ε, ευελιξία στον χρηματοδοτικό τομέα. Μα ανησυχούν λίγο οι ε, προτάσει που έγιναν σε ό,τι αφορά ένα προπολογισμό εξισορρόπηση, ένα balancing budget και από εκεί και μετά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε σε ε, αυτόν τον κανονισμό είναι να δώσουμε περισσότερε δυνατότητε σε ό,τι αφορά κανόνε που βασίζονται σε επιδόσει. Δηλαδή να είμαστε λιγότερο περιοριστικοί και κατά συνέπεια να έχουμε λιγότερο κόστο για του εμπλεκόμενου φορεί και να προωθούμε περισσότερο την καινοτομία. Άρα λοιπόν δεν θέλουμε να επανέλθουμε εδώ σε μια προσέγγιση η οποία είναι περιοριστική σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τι επίγειε υπηρεσίε υποστήριξη και εδώ δηλαδή προσπαθούμε να εισάγουμε κανόνες οι οποίες θα βασίζονται στις επιδόσεις ε, και σε ό,τι αφορά τη δημιουργία νέων ε, επιστοποιητικών για κατηγορίες ε, προσωπικού δεν θεωρούμε πως κάτι τέτοιο έχει ιδιαίτερο νόημα. Πάλι δηλαδή πρόκειται για ένα περιοριστικό κανόνα ο οποίος θα αυξήσει και το σχετικό κόστος. Σε ό,τι αφορά τον διεθνή ρόλο που θα μπορούσε να παίξει η ΆΣΑ προφανώς ε, καλείται να παίξει ένα ε, σημαντικό διεθνή ρόλο, αλλά φυσικά θα πρέπει να παραμείνουμε και εντό των όσων προβλέπει η συνθήκη τη Λισαβόνα σε ό,τι αφορά την εξωτερική εκπροσώπηση. Οπότε θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε ό,τι αφορά την ε, διατύπωση του κειμένου του κανονισμού. Αυτά από την πλευρά μα και προφανώ αναμένουμε με ενδιαφέρον την λεπτομερή συνεργασία που θα έχουμε του επόμενου μήνε μαζί σα. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο, ο κ. Μαρινέσκο, συζητή για μία ακόμα φορά Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς να πω ότι θα δώσω την ίδια σημασία σε όλες τις τροπολογίες και σε όλα τα στοιχεία. Ε, τις, ε, τους χώρους σειράξεων, τις ζώνες σειράξεων, τα drones, οτιδήποτε. Μπορώ να λάβω υπόψη λοιπόν κάθε πρόταση για τη Eurocontrol να πω ένα πράγμα. Δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη μεταξύ της Eurocontrol και του EASA εκτός από αυτό το κομμάτι του κανονισμού για την ε, διαχείριση της και κυκλοφορίας. Η Eurocontrol είναι ο διαχειριστής ε, που έχει ορίσει η Κομισιόν και πληρώνεται γι' αυτό. Δουλεύει και ως φορέας αξιολόγησης της απόδοσης και πληρώνεται γι' αυτό. Έχει οριστεί από την Κομισιόν και μέχρι το 2009 επίσης δούλευε για τη ρύθμιση της ενέργειας κυκλοφορίας. Το 2009 εμείς πήραμε αυτή την αρμοδιότητα από τη Eurocontrol. Δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο υπηρεσιών. Είναι και τα δύο διαφορετικά. Το ένα είναι το ευρωπαϊκό το καθένα έχει τη δική του αρμοδιότητα και όταν υπάρχουν ε, χρήματα για τη, στη συζήτηση, τα λόμπις πάντοτε είναι πολύ ισχυρά. Έτσι λοιπόν, ε, να πω ότι έκανα και μια συνάντηση με τον κύριο Μπέρνερ και τον και του είπα ότι θα πάρω υπόψη κάθε πρόταση, αλλά θέλω γραμμή-γραμμή να βρω τον προϋπολογισμό της Eurocontrol και να δω πού πάνε τα χρήματα από τα τέλη. Αν πάνε στο ρυθμιστικό έργο, να το συζητήσουμε. Κατά την άποψή μου, η πρόταση της Κομισιόν σε αυτόν τον τομέα είναι σωστή. Δεν πήρα πληροφορίες από το Eurocontrol, περιμένω ακόμα. Συγκεκριμένα πράγματα, τις γραμμές του προϋπολογισμού, για να δω πού χρησιμοποιούνται τα χρήματα από τα τέλη. Για τα drones με την κυρία Πρόης ήδη έχουμε ξεκινήσει τη συνεργασία μας και ήδη έχουμε μια ημερομηνία συνάντησης, αλλά έχω ένα πρόβλημα εκείνη την ημέρα. Παρ' όλα αυτά θα το συζητήσουμε αργότερα, όμως ε, όποιος άλλος θέλει μπορεί να έρθει και να συναντηθεί μαζί μας και να οργανώσουμε μαζί τη συνάντηση. Είναι σημαντικό να γίνει η συνάντηση αυτή θα εργαστώ για να προσπαθήσω μέχρι τα τέλη της επόμενης εβδομάδας να έχω συμβαστικές λύσεις που θα στείλω στους ε, συναδέλφους. Μετά τις ε, διακοπές, κάθε εβδομάδα μπορούμε να κάνουμε συνάντηση των σκιωδών. Κάθε εβδομάδα. Όμως χρειάζομαι και μια συνάντηση με την Προεδρία της Σλοβακίας για να ξεκαθαρίσω τι θέλουν να κάνουν. Γιατί εάν, ελπίζω όχι, εάν θέλουν να καθυστερήσουν το θέμα, δεν θεωρώ ότι υπάρχει λόγος βιασύνης και για μας. Μπορεί να βρούμε άλλη ημερομηνία και ή οτιδήποτε τέλος πάντων. Το σημαντικό είναι πρώτα να δούμε ποιες είναι οι προθέσεις. Το θέμα αυτό είναι περίπλοκο, είναι σύνθετο, είναι πολιτικό και τεχνικό ταυτόχρονα και γι' αυτό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Ευχαριστούμε η ποιότητα προέχει της ε, ταχύτητας. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στις ε, διαπραγματεύσεις για τους συμβιβασμούς. Πάμε τώρα στο 6. Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Ο Μάρκος Φέμπερ είναι ο εισηγητής και του δίνω αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, λυπάμαι που έχουμε μόνο 253 τροπολογίες και όχι χίλιες όπως ο συνάδελφος Μαρινέσκου. Δεν έχει να κάνει με τον εισηγητή, ελπίζω. Ίσως ε, στις αεροπορικές υπηρεσίες τα πράγματα πάνε πιο γρήγορα από ό,τι στις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Τέλος πάντων, να σοβαρευτούμε. Χαίρομαι. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Θα ήθελα να σας ζητήσω να φύγετε γρήγορα από την αίθουσα για να μπορούμε να έχουμε ησυχία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 Αν έφυγαν όλοι λοιπόν, μπορείτε να συνεχίσετε. Ευχαριστώ. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι πριν, τώρα έφυγαν τόσοι πολλοί ενδιαφέρον. Τέλο πάντων, για τι ταχυδρομικέ υπηρεσίε έχει να κάνει απλώς εισαγωγικά με μία έκθεση της Κομισιόν, ε, μια οδηγίας που είχαμε ψηφίσει την προηγούμενη ε, θητεία τον Ιανουάριο του 2013. Λοιπόν, ξεκίνησε να ισχύει αυτή η οδηγία. Ε, έπρεπε λοιπόν να υπάρξει αυτή η έκθεση για την εφαρμογή της ε, για να μπορέσουμε να γνωμοδοτήσουμε. Δεν κάνουμε κάποια οδηγία λοιπόν για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες λοιπόν δεν, και αυτή η έκθεση δεν είχαν αυτή την πρόθεση. Να ευχαριστήσω λοιπόν τους Κιώδης ε, που μου έδωσαν τη δυνατότητα να γνωρίζω κι εγώ αυτή την πρόθεση ώστε να συνεργαστούμε σωστά. Προσπάθησα από τις τροπολογίες ε, να βρω μια δομή, να φτιάξω μια διάρθρωση ε, έτσι ώστε να έχουμε 22 συμβαστικές τροπολογίες τελικά, τις οποίες αύριο ελπίζω θα ψηφίσουμε με μεγάλη πλειοψηφία είναι ας πούμε η κοινή θέση, η κοινή μας κατανόηση για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Ε, υπάρχει η καθολική υπηρεσία ως ένα γενικό θέμα εδώ, ένα από τα βασικά στοιχεία λοιπόν της υπαρχής υπηρεσιών, ταχυδρομικών υπηρεσιών. Χαίρομαι που καταφέραμε να εγγράψουμε αυτή την καθολική υποχρέωση υπηρεσίας που πρέπει να τηρείται να μην υπάρχει περιορισμός ή κατάργησή της. Υπήρξαν τροπολογίες σχετικά Ελπίζω λοιπόν ότι η έννοια αυτή της καθολικής υπηρεσίας με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να επανακτήσει το νόημά της, διότι διασφαλίζεται μέσω αυτής ότι όλοι οι πολίτες στην Ευρώπη θα έχουν πρόσβαση στις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Διαπιστώνουμε βέβαια ότι η εφαρμοστική οδηγία των... έχει μεταφερθεί διαφορετικά στα 28 κράτη-μέλη. Έχουμε νέους ανταγωνιστές, έχουμε τις παραδοσιακές ταχυδρομικές υπηρεσίες. Διαπιστώνουμε επίσης ότι η Κομισιόν παίζει λίγο πιο σημαντικό ρόλο από ότι θα μπορούσε σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, δεν είχαμε τόσο μεγάλη διαφοροποίηση σε εθνικό επίπεδο με μικρούς πάροχους κτλ. Για την ευελιξία επίσης εντός της οδηγίας να πω ότι είναι οδηγία, άρα δίνει το πλαίσιο. Αυτή όμως η ευελιξία δεν πρέπει να <clears throat> ξεπεραστεί και αυτό είναι ένα θέμα που συζητήθηκε και βρήκαμε και ένα συμβιβασμό. Η ανεξαρτησία των εθνικών αρχών, ρυθμιστικών αρχών επίσης, είναι ένα αποφασιστικό ζήτημα και η διαλειτουργικότητα έχει υπογραμμιστεί. Ένα σημαντικό θέμα που έχει να κάνει και με την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς. Για τα δέματα επίσης να πω ότι έχουμε μια πολύ ε, συγκεκριμένη πρόταση και χαίρομαι γι' αυτό και με ευχαριστώ τους, ε, τον Πρόεδρο της Επιτροπής γιατί ξέρω ότι πολλές φορές ε, στη διάσκεψη των Προέδρων είναι δύσκολες οι διαπραγματεύσεις. Εγώ ως Αντιπρόεδρος στην ΕΚΟΝ έχω αναλάβει αυτή την θέση πολλές φορές και φαίνεται λοιπόν ότι στο θέμα αυτό δεν χρειάζεται να θέσουμε μια συγκεκριμένη θέση, μπορούμε να έχουμε το δικό μας φάκελο. Επίσης, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που συνεργάστηκαν μαζί μου, οπωσδήποτε τους Σκιώδης. Την περασμένη εβδομάδα χρειάστηκε να αφιερώσουμε πάρα πολύ χρόνο. Δεν είχαμε βέβαια τη δυνατότητα να κρατήσουμε τις αίθουσες περισσότερο. Ε, αλλά είχαμε χρόνο ώστε να μπορέσουμε αύριο να έχουμε ένα καλό κείμενο για να ψηφίσουμε και παρά την ψηφιοποίηση, τα ηλεκτρονικά και όλες τις υπηρεσίες που υπάρχουν, θα, πρέπει, θα συνεχίσουν οι ταχυδρομικές υπηρεσίες να παίζουν σημαντικό ρόλο και θα πρέπει να τις βλέπουμε και ως ένα μέσο επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Ε, βέβαια, ε, φαίνεται ότι η σύγχρονη τεχνολογία τώρα μας δίνει περισσότερες δυνατότητες από ό,τι είχαμε στο παρελθόν, αλλά στο τέλος <clears throat> ε, υπάρχουν ε, οι, όλες οι υπηρεσίες που δίνονται, ακόμα και η καθολική υπηρεσία, είναι σημαντική, υπόψη, που είπα, όπως είπαμε είναι σημαντικό να τηρηθεί, γιατί υπάρχουν πολλές ε, προθεσμίες. Η Κομισιόν λοιπόν θα πάρει τις ιδέες μας και θα τις ε, χρησιμοποιήσει όχι για μια νέα οδηγία, αλλά για την εποπτεία της ε, επί της αγοράς αυτής. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Και πάλι δεν έχουμε χρόνο. Οι σκιώδει έχουν δύο λεπτά και οι υπόλοιποι ένα λεπτό. Λούση Άντερσον. Ευχαριστώ. Όπω είπε και ο συγητή, έχουμε 235 τροπολογίες. Να τονίσω όμω ότι είχαμε και μακροσκελείς νομοδοτήσει από ΙΜΚΟ και ΕΜΒΙ που τονίζουν ακριβώς τη διατομιακή σημασία του κλάδου των, των υπηρεσιών αυτών. Χαιρετίζω λοιπόν αυτή την κοινή δουλειά του εισηγητή και των σκιωδών εισηγητών για την έκθεση αυτή. Για την ομάδα μας πρέπει να διασφαλιστεί η μακρόπνοη βιωσιμότητα αυτών των υπηρεσιών, το οποίο σημαίνει θα πρέπει να διασφαλίσουμε τις υπάρχουσες προδιαγραφές, διατηρώντας βέβαια τις εθνικές και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Οι χώρε μέλη θα πρέπει να έχουν και ευελιξία όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγία. Βέβαια θα πρέπει να προσέξουμε ώστε να μην είναι αντικείμενο αυθαιρεσίας και κατάχρηση αυτή η ευελιξία. Και η τροπολογία 55 σε αυτό αναφέρεται, μιλώντας για θέματα τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο της οδηγίας. Θα θέλαμε λοιπόν να πούμε ότι η πικρικότητα είναι ένα σημαντικό ζήτημα, αλλά επίση εξίσου σημαντικό είναι να μεταφέρεται η νομοθεσία. Οι ταχυδρομικές λοιπόν υπηρεσίε θα πρέπει να διασφαλιστούν με τρόπο που θα διευκολύνει τα δικαιώματα των πολιτών. Οι καταναλωτέ έχουν δικαίωμα σε αυτέ τι υπηρεσίε και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα των καταναλωτών δεν θα παραβιάζονται. Και πράγματι αυτέ οι ταχυδρομικέ υπηρεσίε όπω και η υπόλοιπη νομοθεσία για του καταναλωτέ πολύ συχνά είναι δύσκολο για του καταναλωτέ να γίνει αντιληπτή. Και έχουμε ιδιαίτερα και μια τροπολογία που ζητά διορθωτικούς μηχανισμούς για τους καταναλωτές στο μέλλον, αν κρυθεί απαραίτητο. Επίσης, χαιρετίζουμε την γνωμοδότηση του αδέρφου George Bach. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας τα κοινωνικά ζητήματα και τα ζητήματα απασχόληση. Ξέρουμε ότι η φιλελευθερωποίηση του κλάδου οδήγησε σε συνθήκε εργασία υποδέστερες όπως και σε συνθήκες άσχημες για τις απολαβές και τις αμοιβέ των εργαζομένων. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει κάποια ισότητα, κάτι το οποίο θέλουμε όλοι. Και νομίζω ότι ένας αποτελεσματικός ταχυδρομικός τομέα στην Ευρώπη χρειάζεται μια βιώσιμη ομάδα εργασία ανθρώπων. Και σε αυτό θα πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ζεκή Φώστερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τον μακρόχρόνιο εισηγητή, ο οποίος το αξίζει μετάλλιο. Ξεκίνησε, <laughs> σαν φαίνεται, πριν από δύο ε, αιώνες. Ευχαριστώ, Μάρξ, Πρέπει να πούμε ότι έχει προχωρήσει αυτό το θέμα και αυτές τα χειρονομικές υπηρεσίες, η σημασία τους αναγνωρίζεται πλήρως εδώ. Και στο ECR εμείς θεωρούμε ότι οι τροπολογίες μας βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Ακούσαμε διάφορε ανησυχίε οι οποίε αναφέρθηκαν, οι οποίε έχουν όμως αντιμετωπιστεί και βεβαίω η ομάδα μας θα υπερψηφίσει στο σύνολο της έκθεσης. Είχαμε βέβαια το κύριο ζήτημα εδώ της καθολικής υπηρεσία. Αυτό αναγνωρίζεται τώρα πια σε όλε τι χώρε μέλη. Αναγνωρίζονται βέβαια και οι προκλήσεις, αλλά ξέρουμε ότι η ταχυδρομική υπηρεσία έχει πια αλλάξει είναι αγνώριστη τα τελευταία χρόνια και αυτό το αναγνωρίζουμε βέβαια. Επίσης χαιρετίζουμε την νέα παράγραφο που υπογραμμίζει το θέμα του ανταγωνισμού, της αγοράς και της καινοτομίας στον τομέα. Και μία παράγραφος επίσης με χαροποίησε οι νέες τεχνολογίες και η χρήση των drones για να διευκολύνουμε βέβαια τις υπηρεσίες παράδοσης στις απομονωμένες περιοχές λαμβάνοντας υπόψη βέβαια και ζητήματα ασφάλειας. Ευχαριστώ λοιπόν τον εισηγητή και βεβαίως θα στηρίξουμε την έκθεση αυτή αύριο. Ευχαριστώ. Παύλ ευχαριστώ το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα από την πλευρά μου να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Νομίζω πως ε, ήταν ευχάριστη και αποτελεσματική συνεργασία μαζί του. Και εμεί ε, θέλουμε να υπάρξει μια εύρυθμα λειτουργούσα αγορά για τι τεχνικέ υπηρεσίε ε, για του πολίτες μας, για τους καταναλωτές μας ε, και όχι βέβαια για τους καταναλωτές ε, του 1997 αλλά και τους καταναλωτές του 21ου αιώνα. Ε, και βέβαια αυτό αναγνωρίζεται και στην πρόταση. Τώρα, τι ακριβώς χρειαζόμαστε σήμερα. Χρειαζόμαστε ένα καλό κανονιστικό πλαίσιο το οποίο θα μας θα επιτρέψει την ύπαρξη καλών αποτελεσματικών ταχυδρομικών υπηρεσιών με κάποιο βαθμό ευελιξίας. Και βέβαια θα θέλαμε να υπάρξει μια ανεξάρτητη θέση σε αυτό το πλαίσιο και ισχυρή θέση των εθνικών ε, ρυθμιστικών αρχών. Θέλουμε να αυξηθεί η διαφάνεια στον τομέα στο μέλλον και θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη αποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά τι διασυνοριακέ παραδόσει. Ταυτόχρονα θα θέλαμε να δούμε ένα νέο πλαίσιο το οποίο θα είναι πιο δίκαιο ανάμεσα στου νέου παίκτε στην αγορά ε, και εκείνου που ήδη έχουν εντρεωθεί ε, σε ό,τι αφορά ειδικότερα τα, τους παρόχους Universal Service Obligation. Εκείνο που δεν πρέπει να κάνουμε όμως είναι να παράσχουμε προστατευτισμό. Και αυτό βέβαια αφορά ε, όλη την προσέγγιση της ε, περαιτέρω ανάπτυξης ε, της αγοράς. Δηλαδή όλοι μιλάμε για αυτό, αλλά τελικά κάποιες από τις τροπολογίες ή πολλές από αυτές κατευθύνονται πηγαίνουν προ την αντίθετη κατεύθυνση. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί ούτω ώστε πραγματικά να επιτρέψουμε στην αγορά να αναπτυχθεί. Δύο καταληκτικά σχόλια θα ήθελα να κάνω να υπάρξει, να καταστεί πιο ευανάγνωστο το ε, κείμενο και πιο σαφές, ε, θα πρέπει να περιοριστούμε στις αρμοδιότητές μας. Δηλαδή μερικές φορές υποβάλλουμε ε, τροπολογίες που αφορούν το τομέα της απασχόλησης και ούτω καθεξής, οπότε θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Εμείς θα υπερψηφίσουμε όλες τις συμβαστικές τροπολογίες εκτός από μία και θα προσπαθήσουμε βέβαια να είμαστε πάντοτε θετικοί. Αυτά και περιμένουμε την ψηφοφορία. Μαρία Κίλεν έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ από την πλευρά της ε, κυρίας Κονσάλες που εκπροσωπεί την ε, ΓΟΥΑ. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τον εισηγητή όσο και τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες για την πρόοδο που επιτυχουμε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Όπως διαπιστώσαμε δεν πρόκειται για μια εύκολη ε, έκθεση γιατί οι απόψεις μας σε ό,τι αφορά τις ε, ταχυδρομικές υπηρεσίες και οι απόψεις μας σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της οδηγίας είναι αρκετά διαφορετικές μεταξύ δηλαδή τόσο των πολιτικών ομάδων όσο και μεταξύ των διαφορετικών κρατών μελών. Άρα λοιπόν προσπαθήσαμε από κοινού με τις άλλες ε, ομάδες να βελτιώσουμε το κείμενο για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τις αναφορές που κάνει στη σημασία της λήψης υπόψη των γεωγραφικών και δημογραφικών ιδιαιτεροτήτων και χαρακτηριστικών των επιμέρους κρατομέλων, σε ό,τι αφορά την διασφάλιση της παροχής μακροπρόθεσμων ε, υπηρεσιών αλλά και σε ό,τι αφορά την βελτίωση την ε, βελτίωση των συνθήκων της εργασίας ε, σε αυτό το τομέα, οι οποίες πολύ, συχνά δεν είναι τυπικές συνθήκες εργασίας και σχόνται κάτω από τα πρόβλημα. Κύριε Μαντελέχη, το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η συνάδελφος μου δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα, ζητώ συγγνώμη εκ μέρους της. Πάντως μου δίνει τη χαρά να σας ε, μεταφέρω την απόψή της για την έκθεση. Καταρχάς και εισηγητά συγχαρητήρια για την δουλειά σας. Εμείς έχουμε καταθέσει πολλές τροπολογίες. Καταρχάς αυτές που τονίζουν τις καλύτερες ταχυδρομικές υπηρεσίες παντού. Όχι μόνο στις ε, απομονωμένες περιοχές. Μετά για τους εργαζόμενους. Αυτό είναι ένα θέμα νομίζω που αφορά και τις 22 συμβαστικές προτάσεις από τις οποίες είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχθούμε τις 20. Αυτά από εμά, συγχαρητήρια και πάλι. Die nächste ist Daniela Ayuto. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Συγχαρητήρια στον εισηγητή για τη θαυμάσια δουλειά του. Εμείς θα υποστηρίξουμε αυτή την έκθεση ως εφαρμογή της οδηγίας επειδή λαμβάνει υπόψη τις κάποιες πτυχές που προσπαθήσαμε να επαναφέρουμε με τις τροπολογίες μας. Καταρχάς, η προστασία των διασυνορικών εσωτερικών διασυνολικών μεταφορών, το θέμα της ευελιξίας. Επειδή στην αρχική οδηγία είχε προβλεφθεί αυτή η ευελιξία, τώρα προσπαθήσαμε να περιλάβουμε και το θέμα των απομονωμένων περιοχών, το θέμα της πυκνής κατοίκησης. Για τις μακρινές περιοχές συμφωνούμε. Τώρα για την πυκνότητα κατοίκησης διαφωνούμε και εδώ είχαμε κάποιες αφιβολίες. Για την προστασία των εργαζομένων θα πρέπει βέβαια να είμαστε προσεκτικοί επειδή και εδώ έχουμε ζητήματα κοινωνικού dumping. Να μην ξεχνάμε ότι πολλές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες ιδιωτικού τύπου παρουσιάζουν προβλήματα, είναι προβληματικές όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων για τις νέες τεχνολογίες και τα drones και τη χρήση τους, όπως λέει συνάδελφος Φώστερ. Είμαστε βέβαια υπέρ αυτής της καινοτομίας, όμως να προσέξουμε λίγο το κίνητρο αυτής της τεχνολογίας που πρέπει να βοηθηθεί, αλλά πρέπει να προσέξουμε ώστε να μην στρεβλώσουμε την αγορά. Να προσπαθήσουμε δηλαδή να μην διευκολύνουμε υπερβολικά την χρήση νέων τεχνολογιών εις βάρος αυτών που θέλουν να παράσχουν μια υπηρεσία η οποία θα γίνεται βάση λιγότερο εξελιγμένων τεχνολογιών. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι η σχέση με τους καταναλωτές και που συνδέεται με την βούληση ανάκτησης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Κάνοντας τι, ε, εφαρμόζοντας και υλοποιώντα την αποτελεσματικότητα και την ποιοτική εξυπηρέτηση. Και αυτό είναι βέβαια κάτι που μας βρίσκει και εμά πολύ υπέρ. Ευχαριστώ. Η Μαρίν Καστίνα Νοτιού, η επόμενη μιλήτρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ομάδα μου, όπως γνωρίζετε, την ιδιαίτερη σημασία στην προάσπιση των δημοσίων υπηρεσιών, ιδιαίτερα των ταχυδρομικών. Γι' αυτό ακριβώς είμαστε αντίθετοι με τη μεταρρύθμιση αυτή και τις επιπτώσεις της. Ό,τι και να πει κανεί, σε όλε τι χώρες τη Ένωσης θα έχουμε την πλήρη εξάλληψη των ταχυδρομικών υπηρεσιών καθολικού χαρακτήρα, δηλαδή για όλους, ακόμα και για τι απομονωμένες περιοχές. Οι τροπολογίε που κατέθεσα αγνοήθηκαν στι συμβαστικέ επειδή απλά και μόνο προέρχονταν από την ευρωσκεπτιστική μας ομάδα. Οι μόνες συμβαστικές ε, τροπολογίες ακολουθούν τη δική σας ιδεολογία, την ευρωπαϊκή στική. Μαζί με κάποιες περιτές, θα έλεγα, από κάποιες άλλες ομάδες. Νομίζω ότι είναι ώρα να ανοίξτε τα μάτια, αλλά αυτό δεν ισχύει. Τα κλείσατε περισσότερο. Είναι βλαβερή αυτή η έκθεση. Και μετά η τροπολογία ήταν ακόμα βλαβερότερη. Μετά μη σας φαίνεται λοιπόν παράξενο ότι οι λαοί είναι όλο και πιο εξοργισμένοι στην Ευρώπη και αυτό αξάνεται συνεχώς. Ευχαριστώ. Θα ήθελα από την πλευρά μου και εγώ να εκφράσω την αναγνώριση απέναντι στο έργο που έχει καταβάλει ο Σαλφός Μάρκους ε, Θα ήθελα ε, σε τρία σημεία να επιστήσω την προσοχή με τα οποία ασχολείται και εκείνο στην εκθέση του ε, διατήρηση των υπηρεσιών, των universal υπηρεσιών, δηλαδή καμία τροποποίησή τους ή περιορισμός τους, πράγμα το οποίο είναι και για μένα πολύ σημαντικό. Μετά δεύτερο σημείο είναι ο ρόλος ε, των ε, κανονιστικών αρχών, δηλαδή στο πλαίσιο της απελευθέρωσης των αγορών, είναι πάρα πολύ σημαντικό οι ε, κανονιστικές αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να παραμείνουν ισχυρές και πάνω απ' όλα ανεξάρτητες. Και το τρίτο σημείο είναι οι κοινωνικές πτυχές, η κοινωνική διάσταση, αν θέλετε, για τις οποίες βέβαια χαίρομαι ως εκπρόσωπος της πολιτικής μου ομάδας στην ε, Επιτροπή Απασχόλησης για το γεγονός ότι έχουν ληφθεί υπόψη πάρα πολλές από αυτές τις ε, κοινωνικέ ε, πτυχές υπόψη στην έκθεση. Ευχαριστώ. Ισαπέλα Ντεμόντ, έχετε το λόγο. Πρώτα ευχαριστώ. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή και του κοιόδης για τη δουλειά τους. Να υπογραμμίσω μόνο κάτι από τη δικιά μου την πλευρά. Το γεγονό ότι έχουμε μείωση της κύριας υπηρεσίας, δηλαδή η παράδοση των επιστολών, αυτό από μόνο του θα πρέπει να μας οδηγήσει μια διαφορετική αξιολόγηση σε σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή, ποια είναι η κύρια δραστηριότητα, η οποία πια είναι σχεδόν περιθωριακή σε σχέση με άλλες υπηρεσίες, οι οποίες είναι συμπληρωματικές αλλά οικονομικά πιο σημαντικές για αυτούς που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Ταυτόχρονα είναι σαφές ότι η ψηφιοποίηση επηρεάζει σημαντικά τους καταναλωτές και τη συμπεριφορά τους. Οπότε θα πρέπει να συνδυάσουμε τη βιωσιμότητα αυτών των δραστηριοτήτων με τη διατήρηση μιας υπηρεσίας η οποία είναι καθολικού χαρακτήρα και αφορά το δικαίωμα όλων να απολαμβάνουν αυτές τις υπηρεσίες. Το άρθρο λοιπόν 54, κατά την άποψή μου, μπορεί, και αυτό αναφέρεται στις συμβαστικές προτάσεις, να αποτελέσει ένα καλό συμβασμό. Δηλαδή, όσο προχωράμε στην ψηφιοποίηση των απομακρυσμένων περιοχών, θα μπορούσαμε ταυτόχρονα εξίσου να περάσουμε σε μεγαλύτερη ευελιξία. Επίσης, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το γεγονό ότι οι χώρες μέλη παρέχουν διαφορετικές υπηρεσίε, οπότε και εδώ πρέπει να υπάρχει κάποια διαφορετική φύση ευελιξία, η οποία θα αφορά μόνο τι χώρες μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα ο και εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία, λέει ο πρόεδρο. Η κυρία, ζητώ συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να σχολιάσω. Ευχαριστώ πολύ για τη δουλειά του Κοινοβουλίου σε αυτή την έκθεση βίας πρωτοβουλίας. Όπως ε, υπόθηκε Πέρυσι, στην έκθεση για την εφαρμογή της Κομισιόν φαίνεται ότι οι ταχυδρομικές υπηρεσίες ε, αυτή τη στιγμή βιώνουν μια θεμελιώδη αναδιάρθρωση, όπως ας πούμε μέσω της ψηφιοποίησης. Είπαμε ότι δεν, είδαμε ότι δεν υπάρχει ανάγκη να αλλάξουμε την ε, οδηγία αυτή τη στιγμή, γιατί είναι οδηγία πλαίσιο, υπάρχει ευελιξία στον τρόπο ερμηνείας της ε, από τα κράτη-μέλη. Ταυτόχρονα όμως, λόγω της αλλαγής στην αγορά, χρειάζεται μια καλύτερη παρακολούθηση του πώς εξελίσσονται οι όγκοι των πακέτων και των επιστολών. Σύμφωνα με τις στατιστικές που δημοσίευσε η Κομισιόν στην ιστοσελίδα της, υπήρχε μεγάλη αλλαγή. Ε, υπόθηκαν πολλά για τα πακέτα, για τα δέματα για την, μετά από την πρόταση για καθορι, ε, κανονισμό σχετικά με τις διασυνοριακές υπηρεσίες που εγκρίθηκε το Μάιο. Χαιρετίζουμε αυτά που υπόθηκαν για αυτό το θέμα. Επίσης, συμφωνούμε ότι η αγορά και ο ανταγωνισμός ε, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο γιατί κινητοποιούν την καινοτομία και αυτό ήταν και στον χάρτη των οδικό της Κομισιόν το 2013 για τα δέματα που είχε να κάνει με τον εντοπισμό του στην καθολική υπηρεσία, τα διάφορα προγράμματα και θέλουμε να προχωρήσουμε θέματα όπως η τυποποίηση μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης και θα γίνει περισσότερη συζήτηση για τα διασυνοριακά πακέτα δέματα. Επίσης, για τις ρυθμιστικές αρχές να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να είναι ανεξάρτητες. Έχουμε την ομάδα των ε, ρυθμιστικών αρχών για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που ιδρύθηκε το 2010 και έχει αναλάβει πολύ σημαντικό έργο συντονισμού ε, αλλά και μία πρόσφατη δουλειά που έκανε ήταν το εργαστήριο στη Σόφια σχετικά με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Και αυτό το χαιρετίζουμε. Επίσης αναφέρθηκε η εργασιακή διάσταση που είναι πολύ σημαντική. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής ε, Απασχόλησης. Σύμφωνα με την γνωμοδότηση, τα κράτη-μέλη έχουν ευελιξία ως προς τις εργασιακές ε, συνθήκες, όμως ε, αυτές αλλάζουν από ό,τι φαίνεται και γι' αυτό ελπίζουμε ότι ο κανονισμός για τις διασυνοριακές υπηρεσίες των πακέτων θα βελτιώσει την παρακολούθηση ε, των υπηρεσιών και των εργασιακών συνθήκων σε όλη την Ευρώπη. Ευχαριστούμε πολύ για τη δουλειά σας. Ευχαριστώ τώρα. Έχει το λόγο ο εισηγητής. Ευχαριστώ πολύ. Προσπάθησα να φτιάξω έναν συμβιβασμό παίρνοντας ε, το ζουμί από τις τροπολογίες ε, χωρίς να λαμβάνω υπόψη βέβαια και τους στόχους ε, της οδηγίας. Είναι καλό λοιπόν που θα μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε και αυτό. Να πω λοιπόν ότι η ιδέα της καθολικής υπηρεσίας χρησιμοποιείται ξεκάθαρα στις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Αυτό στην ουσία είναι κάτι διαφορετικό από την υποχρέωση δημόσιας υπηρεσίας. Επίσης, ε, μέσα στα πλαίσια αυτής της καθολικής ε, ε, υπηρεσίας έχουμε ανοίξει χώρο για τον ανταγωνισμό. Είχαμε, λοιπόν... είδαμε λοιπόν ότι στην οδηγία και στην έκθεση δεν υπάρχει ούτε λέξη για ιδιωτικοποίηση ή κάτι τέτοιο και επίσης κάποιοι συνάδελφοι ίσως να έχουν κάποια διαφορετική θεώρηση για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Αύριο, ε, βέβαια, όταν θα έχουμε τη μεγάλη πλειοψηφία, θα καταλάβουν ότι τα πράγματα είναι αλλιώς και χαίρομαι ιδιαίτερα που τουλάχιστον σε αυτή την Επιτροπή υπάρχει βασικά σύμπνοια. Ελπίζω λοιπόν ότι ε, αυτό σημαίνει ότι και τα νομοθετικά μέτρα που έχουμε μπροστά μας, όπως ας πούμε αυτά για τα δέματα θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε θέματα πιο γενικά με επικοδομητικό τρόπο. Ευχαριστώ λοιπόν για το επικοδομητικό πνεύμα και ελπίζω ότι αύριο θα έχουμε και την θετική κατάληξη. Ευχαριστώ πολύ. Να πω ότι αύριο ψηφίζουμε αυτή την έκθεση. Περνάμε στο επόμενο σημείο προπολογισμό 2017. Συγγήτρια είναι η κυρία Ισάβελα Τελμότο και τη δίνω κατευθείαν το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Σύντομα να σας παρουσιάσω το περιεχόμενο που περιλαμβάνει και τις μεταφορές αλλά και τον τουρισμό. Για τις μεταφορές. Κυρίως υπογράμμισα ότι εδώ δεν έχουμε πετύχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και αυτό έχει λεχθεί επανειλημμένο στην Επιτροπή μας. Οπότε οι περικοπές αυτών των ταμείων δεν θα έπρεπε να είχαν λάβει χώρα. Θα πρέπει λοιπόν να αποκατασταθούν τα ταμεία αυτά και να καλύπτουν μεταφορές με ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Βλέπουμε επίση να υπάρχει μια μετατόπιση των μεταφορών προ τι οδικέ μεταφορέ. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο θα πρέπει να υπάρξει μια κατάλληλη χρηματοδότηση κατάλληλη και για θαλάσσιες αρτηρίες έχουμε τον Ευρωπαϊκό Συνδρομικό Οργανισμό. Ζητάμε να υπάρχει και η κατάλληλη χρηματοδότηση για να διαδραματίσει το ρόλο που του αρμόζει. Επίσης έχουμε και ένα περιβαλλοντικό ζήτημα, το ζήτημα της ε, βιωσιμότητας, που είναι και οικονομικό αλλά και περιβαλλοντικό, ώστε δηλαδή να υπάρχουν στόχοι οι οποίοι απορρέουν από την COP21, πέρα δηλαδή από την αποτελεσματική διαχείριση της ε, ενουσιακής επιμελητίας. Υπάρχει επίσης και το ζήτημα του τουρισμού που ακολουθεί κάπως τη γραμμή του ψηφίσματος που εθετήσαμε στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου όπου ζητάμε την θέσπιση μιας συγκεκριμένης γραμμής στον προπολογισμό για τον τουρισμό και για λόγους διαφάνειας. Να δούμε δηλαδή επιτέλους πόσο θέλουμε να επενδύσουμε σε αυτό το σημαντικό κλάδο της ευρωπαϊκής οικονομίας. Εδώ για το γλωσσικό θέμα, για τους οδηγούς, να συγχαρώ την Κομισιόν. Ξέρω ότι ξεκίνησε αυτή η δουλειά και ήδη έχει δώσει καρπούς. Πριν από λίγο Μιλήσαμε για διάφορες ε, απομονωμένες, απομακρυσμένες, παράκτης, φρονές περιοχές κτλ. Και αυτό αναφέρεται εδώ, σε αυτή τη γνωμοδότηση, γιατί στην ουσία αποτελεί ένα πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή η προώθηση του πλούτου αυτών των πιο ασθενών <laughs> περιοχών πρέπει να οδηγήσει και στην αναδιανομή των κονδυλίων, ώστε να βοηθήσουμε αυτές τις περιοχές. Και τέλος, η διευκόλυνση της πρόσβασης στις τουριστικές δομές των ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα. Ξέρουμε ότι αυτό είναι σημαντικό πρόβλημα στον τομέα του τουρισμού και θα πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά. Αυτά είναι κάποιες έτσι γενικές γραμμές. Βέβαια είμαι στη διάθεσή σας αν θέλετε περισσότερες ε, λεπτομέρειες ή διευκρινήσεις. Ο κ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την έκθεση. Καλύπτει τα θέματα αρμοδιότητάς μας ως Επιτροπής. Να πω ότι ο προπολογισμός του 17 είναι πολύ σημαντικός. Γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα που θα πρέπει να ρυθμίσει η Κομισιόν, η οποία αναζητεί τα χρήματα. Ψάχνει λοιπόν στον προπολογισμό επειδή οι χώρες μέλη δεν είναι διατεθειμένες να συνεισφέρουν περισσότερα. Ξέρουμε ότι οι συνεισφορές είναι χαμηλότερες από αυτές του 16. Είχαμε γύρω σε 6% περικοπές στον προπολογισμό. Δεν είναι καλό αυτό, οπότε θα πρέπει να προσπίσουμε τα κονδύλια για τις μεταφορές και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα πρέπει να ζητήσουμε ξεκάθαρα να συμπληρωθούν τα κονδύλια για τις εσωτερικές γραμμές των μεταφορών της Κομισιόν και ό,τι λείπει να το πάρουν από τα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Και μετά να ψάξουν αλλού για το πώς θα τα καλύψουν αυτά. Αλλά όπως είδαμε και στο Στρασβούργο, έχουν μόνο ένα δις και τα projects στο, στο που συζητάμε είναι προγράμματα μακρόπνοα Νομίζω ότι του χρόνου κιόλα έχουμε τι προθεσμίε, το οποίο σημαίνει ότι μέχρι του χρόνου θα πρέπει να γνωρίζουμε τι γίνεται. Αυτή είναι λοιπόν η πρότασή μου κιόλα. Να δούμε τι γίνεται με αυτά τα ζητήματα, να δούμε τι γίνεται με τι εσωτερικέ πλούτε οδού, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με όλα αυτά και το TMS επίσης. Τη μετατόπιση προς τις συνδρομικές μεταφορές να δούμε τι γίνεται εκεί με τη χρηματοδότηση από τις οδικές της συνδρομικές και το CSR βέβαια και αυτό είναι το πιο σημαντικό νομίζω εξάλλου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Παπαντελίσκα. Ευχαριστώ. Ε, λυπάμαι πρέπει να φύγω. Δεν έχω χρόνο να μιλήσω. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. η κυρία Κερμαντιλή. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ε, τότε να μιλήσω παραπάνω, αφού θα φύγει ο συνάδελφο. Α, μια χαρά. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, γιατί σε γενικέ γραμμές να πω ότι συμφωνώ μαζί της. Η ομάδα μου θεωρεί ότι αυτά που γράφεται είναι σωστά. Έχω μόνο κάποιες διευκρινήσεις. Καταρχάς να τονίσω κάτι του χρόνου το 2017 θα είμαστε ένα έτος μετά το δημοψήφισμα. Εγώ θεωρώ ότι τότε ακριβώ θα πρέπει να τονίσουμε το γεγονό ότι εμεί θέλουμε να υπάρχει ένα πραγματικό προπολογισμό συμφιλιωτικό. Δηλαδή σήμερα είμαστε υπερχρεωμένοι να έχουμε τέλο πάντων μεταφορά αυτή τη δημοσιονομική προσπάθεια από την Κομισιόν που γίνεται ει βάρο συνήθω των δομών των μεταφορών. Μπορούμε όμω να κάνουμε έναν συμβασμό γιατί οι μεταφορές είναι κάτι το καθημερινό ως φαινόμενο. Οπότε τι μπορούμε να κάνουμε εδώ. Μετά. Για το τι. Εμείς είμαστε υπέρ της ανάπτυξης των διασυνοριακών μεταφορών. Θέλουμε όμως τα μεγάλα project να συνοδεύονται και από μικρότερα. Αυτό που είπατε το άκουσα προσεκτικά, αλλά θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σοβαρά. Για τον προπολογισμό. Έχουμε τα κονδύλια τα οποία θα πάνε να τροφοδοτήσουν το Ταμείο Juncker. Εκεί δεν έχουμε αντίρρηση. Έχουμε όμως αντίρρηση για το εξής τα μισά προγράμματα Juncker είναι υποδομών ή διεύρυνση αυτοκινητοδρόμων. Κάτι το οποίο είναι αντίθετο με το στόχο της Κομισιόν που λέει ότι θα πρέπει να αποανθρακοποιήσουμε τι μεταφορές. Αν λοιπόν με αυτό το στρατηγικό ταμείο επενδύσεων η Κομισιόν δεν θέλει να κάνει πολλαπλούς τρόπους μεταφορών, ούτε βιώσιμες μορφές μεταφορών, ε, μεταφορών ούτε νέες τεχνολογίες κτλ. Τότε αυτός ο προπολογισμό είναι λίγο προβληματικός. Έχουμε και τα θέματα προστασίας των επιβατών. Αυτά είναι λοιπόν ζητήματα τα οποία θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Κάτι άλλο ενδιαφέρον στην εκθεσή σας είναι ότι επιτέλους βλέπουμε να γίνεται μια προσπάθεια ανάπτυξη του, του σιδηροδρόμου. Εδώ θα πρέπει να επιμείνουμε γιατί έχουν υποεπενδύσει οι χώρε μέλη στην διατήρηση και συντήρηση των σιδηροδρομικών υποδομών. Θα πρέπει να επαναεπενδύσουμε στα σιδηροδρομικά συστήματα τα οποία σημαντικά πανευρωπαϊκά. Και στο τέταρτο συνολικό πακέτο έχουμε τον τεχνολογικό πυλώνα. Αν θέλουμε λοιπόν να κάνουμε εξοικονομήσεις μακροχρόνιες, μέσω τεχνολογίας θα πρέπει καταρχάς να κάνουμε επενδύσει για την ενορμόνιση των συστημάτων ασφάλειας και της διαλειτουργικότητας του υλικού, κάτι το οποίο απαιτεί μια σοβαρή προσπάθεια οικονομική, στην οποία θα πρέπει να συνεισφέρει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι. Αυτό είναι σημαντικό. Να έχουμε λοιπόν υπόψη μας ότι οι μορφές αυτών, των μεταφορών δεν θα μεταφερθούν αυτόματα στο σιδηρόδρομο. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την ήπια μετακίνηση, με το τρένο, ήπιες μεταφορές κλπ. Οπότε σε αυτό το σημείο θα πρέπει να ενισχύσετε κάπως τα λεγόμενα της έκθεσής σας. Και κατά λίγο πρόεδρε, θα πρέπει να επιμείνουμε στο θέμα των νέων τεχνολογιών. Υπάρχει μια νέα γενιά μεταφορέων και μεταφορών που είναι η κινητικότητα του αύριο, που είναι έξυπνη, που είναι ευφυής και που πραγματικά αποτελεί μια εναλλακτική λύση στη χρήση του αυτοκινήτου. Και το ερώτημα είναι πώς μπορούμε πραγματικά να βοηθήσουμε αυτούς τους νέους εφευρέτες της αυριανής κινητικότητας ώστε να αναδειχθούν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Danke sehr. Die nächste ist Daniela Ευχαριστώ. Και μετά η Μαρίν Κριστίνα Νότου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, συμμερίζομαι την άποψη που λέει ότι το έτσι είναι ένα ταμείο στήρο και ότι ε, οι μηχανισμοί για τη διαλειτουργικότητα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την χρηματοδότησή του. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση ε, λέγεται ότι πρέπει να ευνοηθούν οι θαλάσσιες μεταφορές σε σχέση με τις σιδηροδρομικές, όμως ε, βάσει του τέταρτου πακέτου για τις σιδηροδρομικές μεταφορές που θα ε, τεθεί σε εφαρμογή τον, το φθινόπωρο. Όμως, οι οδικές μεταφορές είναι πάρα πολύ ε, πιο ανεπτυγμένες και έχουμε περάσει από τις ε, ράγες ε, στο δρόμο, κάτι που δημιουργεί και κοινωνικό dumping. Χρησιμοποιείται λοιπόν το προσωπικό με τρόπο που δεν πρέπει και πρέπει να επαναεξισορροπήσουμε την κατάσταση. Είπα όλα όσα ε, πίστευα στη γνωμοδότηση για την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και όλα τα άλλα που αφορούν ε, το ε, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θαλασσίων Μεταφορών. Βέβαια, απορρίφθηκαν οι εκθέσεις μου και επειδή ήμουν η μόνη εισηγήτρια, παρά να χαρούμε ε, παρά το γεγονός ότι χαρήκαμε τελικά για την έγκριση της ε, εισήγησης ε, αυτής, όταν την έκθεση πήρατε εσείς κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ η κυρία Ντομινίκ Λεκλέ. Ο κύριος Ντομινίκ Λεκλέ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω εκ μέρους του συντρόφου που έφυγε πρόωρα. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την έκθεσή της. Ε, θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, ικανοποιητική και πλήρης. Εγώ ήθελα να πάω λίγο πέρα από τις γενικές παρατηρήσεις που εντάξει πάντοτε αξίζει να επαναλαμβάνουμε, αλλά να κάνω πιο συγκεκριμένες παρατηρήσεις για τον προϋπολογισμό. Λέει η εισηγήτρια ότι το έτσι δεν έχει δώσει τα αποτελέσματα που θα θέλαμε. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε, γιατί το ταμείο αυτό προβλέπεται για τρία έτη. Όμως η ανάπτυξη μακροπρόθεσμων ε, επενδύσεων δεν μπορεί να αξιολογηθεί μέσα στους τρεις πρώτους μήνες. Έτσι λοιπόν τα πρώτα αποτελέσματα δεν δείχνουν ακριβώς αν έχουμε πάει στη σωστή κατεύθυνση. Δεν μπορούμε επίσης να πούμε ότι ε, δεν είχαμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Φαίνεται ότι, όπως είπανε και όλοι εδώ, ένα κομμάτι του ταμείου ήταν από τα τέλη που είχε να κάνει με τις επιχορηγήσεις ε, και αυτό μας έκανε να έχουμε κάποιες ελπίδες οι οποίες τελικά διαψεύστηκαν, όμως τα δύο έπρεπε να ε, λειτουργήσουν ταυτόχρονα. Άρα υπάρχει ανάγκη να υπάρχει ένας μηχανισμός bundling, ο οποίος ε, θα, ε, θα εφαρμοστεί και σε αυτό το θέμα. Και το λέμε τώρα, αρνούμενοι μια, ένα νέο τέλος. αυτό που προτείνει η Κομισιόν όχι ως άμεσο τέλος, αλλά ως τέλος σε κάποια χρηματοπιστωτικά εργαλεία, τα οποία θεωρώ απαράδεκτο. Ε, χαιρόμαστε επίσης για το τέταρτο πακέτο των σιδηροδρομικών μεταφορών. Δεν έχουμε καν ψηφίσει γι' αυτό, πώς συγχαίρουμε, τέλος πάντων, για το τέταρτο πακέτο. Για τα τεχνικά σημεία να πω ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Μια άλλη παρατήρηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι πρέπει να επανέλθουμε στο προϋπολογισμό αυτό καθεαυτό και να κοιτάξουμε το κεφαλαιο 1α το οποίο πρέπει να εξισορροπήσει κάποια πράγματα τα οποία περιμένουμε από τον προϋπολογισμό και να μην κοιτάμε λίγο περισσότερο τον προσανατολισμό γιατί και, αυτοί παίζουν, και αυτές οι παρατηρήσεις παίζουν ρόλο αλλά δεν είναι συγκεκριμένες για τον προϋπολογισμό. Επίσης, να πω για το ρόλο της ε, ε, Κομισιόν για το Ταμείο, ότι ε, τα περιθώρια, η δυνατότητα να μιλήσουμε για ευελιξία σε αυτόν τον προϋπολογισμό είναι πράγματα που πρέπει να θέσουμε επιτάπητος. Πρέπει το Ταμείο αυτό έτσι, να αυξήσει λίγο την οπτική του σε αυτό το θέμα, διότι ε, στο μέλλον, όχι το 2017, αλλά το 2018 ή 19 ή 20, θα χρειαστεί να δούμε το θέμα πιο συγκεκριμένα και το 2017 θα είναι η τελευταία χρονιά που η Βρετανία θα δίνει τόσο γενναιόδρα τη συνεισφορά της στον προϋπολογισμό μας. Ευχαριστώ. Ρόμπερτ Ζήλ. Ευχαριστώ, συγγνώμη που άργησα. Εκ μέρους του ECR θέλω να πω και εγώ μερικά πράγματα. Καταρχάς, ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για αυτή την έκθεση. Το ECR πάντοτε υποστήριζε τις προτάσεις για τον προϋπολογισμό, εφόσον είναι ρεαλιστικές και συγκεκριμένες. Συμφωνούμε για τις υποδομές ως ραχοκοκαλιά της ενιαίας αγοράς και της ελευθερίας μετακίνησης αγαθών και προσώπων. Έτσι λοιπόν ο προϋπολογισμός πρέπει να διανέμεται σωστά ώστε να επιτυχάνουμε αυτούς τους στόχους ε, για τα δίκτυα για, ε, ως το 2030 και τα ολοκληρωμένα δίκτυα στο 2050 όπως αναμέναμε τα αποτελέσματα σε επίπεδο πολιτικής μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ικανοποιητικά. Η ιδιωτική χρηματοδότηση από τα έτσι δεν πηγαίνει στην κατεύθυνση που εμείς θεωρούσαμε ως ε, προτεραιότητα, ας πούμε τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Δίνονται χρήματα σε πιο παραδοσιακά project που όμως δεν είναι περιβαλλοντικά, φιλικά ή μακροπρόθεσμα ε, θα μπορούσαν να αλλάξουν τις πολιτικές. Επίσης, οι προτεραιότητες του Connecting Europe δεν είναι ίδιες με αυτές του έτσι, άρα ε, το έτσι έχει και κάποια γεωγραφική κατανομή. Εκεί που υπάρχει υψηλότερο ΑΕΠ κατά κεφαλήν ή μεγαλύτερη πυκνότητα πληθυσμού, μεγαλύτερο εμπόριο, υπάρχουν περισσότερα project. Και αυτό δεν είναι μεγάλη έκπληξη και σε κάποιες περιπτώσεις, με λίγο χιούμορ ας πούμε να πούμε, ή μια φήμη ε, λέει ότι τα project αυτά στην ουσία ε, αντικατοπτρίζουν τις ε, επισκέψεις του Πρόεδρου της Κομισιόν τους τελευταίους 18 μήνες. Για την Επιτροπή λοιπόν Μεταφορών θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, υποστηρίξουμε την πρόταση του εισηγητή σχετικά με το ότι οι περικοπές του Connecting Europe ε, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως κονδύλια για το έτσι. Γιατί ε, αυτό θα ήταν επικίνδυνο όχι μόνο για την ενδιάμεση αναθεώρηση, αλλά και για τη βασική μέθοδο χρηματοδότησης των μακρόπνων και μεγάλης κλίμακας επενδυτικών project τα επόμενα τις επόμενες δεκαετίες θα έλεγα. Και αυτή είναι μεγάλη πρόκληση για την Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Ο Βιμ Βαντεκάμ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αντίθετα προς την Μαντέλη, εγώ θεωρώ πως, πως ε, η κυρία Τεμόντε έχει ε, συντάξει μία ένα πολύ καλό κείμενο, το οποίο είναι δηλαδή καλά δομημένο, ε, είναι λιτό, ε, δεν έχει πάρα πολλά, αλλά από εκεί και μετά, σε, ό,τι αφορά τα, το ΣΕΦ και το ΕΦΣΥ, ε, προφανώς η Επιτροπή θέλει ε, να λάβει πίσω τα χρήματά της και ε, οι συνάδελφοι Μαρινέσκου ήδη του ανέφεραν, ότι δηλαδή θέλουν τα, τα, τα χρήματα αυτά του ΣΕΦ δεν ξέρω κατά πόσο κάτι τέτοιο θα είχε νόημα. Δηλαδή από τη μία λούμε κάποιο κοντήλι από το ΕΦΣΙ και από την άλλη θα χάσουμε κάτι με όλη αυτή τη διαδικασία. Οπότε ε, το να λέμε ότι το ΕΦΣΙ δεν έχει επιφέρει τα αποτελέσματα που θέλαμε σε ό,τι αφορά τις υποδομές ε, είναι λίγο πρόημο. Δηλαδή ε, δεν ξέρουμε ακόμα αν πραγματικά δεν έχει επιτευχθεί πρόοδο. Μετά σε ό,τι αφορά το άρθρο 4, νομίζω πως, ε, το σημείο 4, νομίζω πως πάει λίγο μακριά εδώ η διατύπωση. Ουσιαστικά δηλαδή λέει ότι ότι θα πρέπει να διευρυνθεί περαιτέρω αυτός ο, ο κλάδος της ε, ε εσωτερικής θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να τροποποιήσουμε αυτή την πρόταση, να είναι πιο σαφή δηλαδή και να μην εκφράσει με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Εγώ ήμουνα στην Πρατισλάβα χθε ε, και είχα βρεθεί εκεί πριν από 33, ε, 33 ε, χρόνια και από το Ιγκελ που πηγαίναμε προ την Πρατισλάβα και κάθε φορά κάθε, πήγαμε με το καρδιά και κάθε 5 λεπτά έπρεπε να προσέχουμε γιατί πέρναγαν ε, κάποια μεγάλα πλοία και κινδυνεύαν από τα κύματα τους. Ε, μετά άλλη φορά βρέθηκα στο Δούναβι και είδα ε, ε, να περνάνε για παράδειγμα πάρα πολύ λίγα πλοία. δηλαδή είδαμε σε κάποιε ε, οδού εσωτερική ναυσιπλοεία ε, να υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αύξηση τη κυκλοφορία, ενώ σε άλλε να έχει μειωθεί πάρα πολύ. Άρα λοιπόν θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ναι, θα υπάρχει ναυσιπλοεία, από την άλλη πλευρά όμω θα υπάρχει και περιβαλλοντική προστασία και θα υπάρχουν και όρια σε ό,τι αφορά τι εκπομπέ στον τομέα. Οπότε ε, ίσως με κάποια σωστά διατυπωμένη τροπολογία θα μπορούσαμε να το επιτύχουμε, να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Ναι, νομίζω ο πρότυπο δεν θα πρέπει πια να κάθεστε σε καγιάκ. Να μην κάνετε άλλο. Ε, εντάξει, ναι, αν ήμουν τόσο νέο, λέει ο πρόεδρο, όπω εσεί, ε, δεν θα έκανα καγιάκ. Αλλά, εν περιπτώσει, να δώσουμε τώρα το λόγο στην Επιτροπή. Κάσμιρ Τσακ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Καταρχήν θα θέλαμε να σας ε, ευχαριστήσουμε για την συνεχή υποστήριξη που μας παρήχατε σε ό,τι αφορά τις ε, πολιτικές ε, μεταφορών και ε, τον προπολογισμό αυτού του τομέα πολιτικής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης την εισηγήτρια Ντεμόντε για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης το οποίο αναλύσαμε προσεκτικά. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι αυτός ο προπολογισμός δίνει στην Επιτροπή ένα πολύ καλό εργαλείο για την εφαρμογή της πολιτικής στο τομέα των μεταφορών για να δώσει έναυσμα στην ανάπτυξη και ε, στην δημιουργία θέσεων εργασίας από τα 3,7 δισεκατομμύρια ε, σε μέρες υποχρεώσεων που έχουν επενδυθεί στις μεταφορές, το 3,2 δισεκατομμύρια, δηλαδή 86% ε, κατευθύνονται προς τις μεταφορές. Και νομίζω πως ε, τα σημεία τα οποία αναφέρεται σε ό,τι αφορά δηλαδή τις οδούς, τις συγκεκριμένες οδούς για τα οχήματα εσωτερικής ναυσιπλοίας και εσωτερικής, να πω ότι οι, στις διαδικασίες για την εκδήλωση ενδιαφέροντος δώσαμε χρηματοδότηση για 80 project με συνολική ε, χρηματοδότηση ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων. Επίσης εκφράστηκαν κάποιες ανησυχίες σε ό,τι αφορά την ΕΦΣΗ. Η ΕΦΣΗ έχει να παίξει το δικό της ρόλο και 17 project τα οποία έχουν ε, ήδη εγκριθεί λειτουργεί πολύ καλά. 12 από αυτά τα project έχουν ήδη υπογραφεί και τα οποία ε, αντιστοιχούν σε 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ και οδηγούν στη δημιουργία 60.000 θέσεων εργασία. Αν λοιπόν συγκρίνουμε ε, την επένδυση των 8,5 δισεκατομμυρίων της ΕΦΣΙ με τα 2,2 ε, ε, με βάση, αν ε, ε, αφαιρέσουμε από τα 8,5 δισεκατομμύρια τα 2,2 δισεκατομμύρια που είχα, έπρεπε να έχουν επενδυθεί στον άλλο τομέα, θα μείνουμε πάλι με 6 δισεκατομμύρια ως τελική επένδυση από την πλευρά της ΕΕ. Ε, τώρα, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον σχετικό τομέα έχει αυξηθεί στα 30 εκατομμύρια ευρώ, σε σύγκριση με τα 26 εκατομμύρια με συμπληρωματικές 16 θέσεις εργασίας, πράγμα το οποίο δείχνει ότι αναγνωρίζεται η σημασία του τομέα, του τομέα της ναυσιπλοείας. Έχουμε 263 άτομα και έχουμε 40% αύξηση του σχετικού προπολογισμού σε σύγκριση με το 2016, το νέο δηλαδή σχέδιο προπολογισμού του 2017. Η σχετική αρχή θα έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει σχετικέ ε, πολιτικέ ε, που, ε, που έχουν συμφωνηθεί και στο πλαίσιο του νέου, της νέας συμφωνίας για την άκτο και συνοριοφυλακή. Επίσης, έχουμε αντίστοιχη αύξηση σχετική υπηρεσία κατά το 20% του προσωπικού. Άρα λοιπόν εδώ βλέπετε μια σύντομη σύνυψη σύνοψη των όσων έχουν συμβεί στο επίπεδο του προπολογισμού και βέβαια από εκεί και μετά ε, είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν ερωτήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και ο λόγος θα πάλι τώρα στην ε, κυρία Ντεμόντε την εισηγητρία μας. Πρώτα ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω καταρχάς όλους τους συναδέλφους για τη σημαντική του συμβολή εγώ από την μεριά μου έχω κάθε διάθεση να δεχτώ προτάσεις για τις τροπολογίες, ενδεχομένω και ακριβέστερες παρατηρήσεις για το ίδιο τον προπολογισμό. Και θα ήθελα να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις ή παρατηρήσεις. Αυτός ο συμβασμός, η συμφιλίωση που πρέπει να κάνουμε στην Ευρώπη, νομίζω ότι έχει ως πρωταγωνιστές τις υποδομές αυτό δηλαδή που συνδέει τις διάφορες χώρες μέλη. Διάδρομοι, συνδέσμοι που λείπουν, κρίκοι που λείπουν, όπως είπαμε προηγουμένως. Αυτό συνδέεται με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, γιατί όταν, βελτιώνονται οι μεταφορές, βελτιώνονται και οι συνθήκε ζωής και εργασίας των ε, πολιτών. Για το σχέδιο Juncker, νομίζω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε το γεγονός ότι είναι δύσκολο να βρούμε μόχλευση για τις υποδομές. Και αυτό είναι τώρα το πρόβλημα τη στιγμή που έχουμε περικοπές από συγκεκριμένα ταμεία. Ταμεία που απέβλεπαν στην διευκόλυνση των υποδομών και αφορούσαν τον σεδρομικό τομέα, αυτόν δηλαδή που ρηπαίνει λιγότερο. Και μια και μιλάμε για το περιβάλλον, όπω έγραψα, μια σημαντική πτυχή είναι η καινοτομία που ισχύει και για τα αναλλακτικά καύσιμα. Και τέλος, για την εσωτερική ναυσιπλοεία, ευχαριστώ να, διατυ... να αλλάξω τη διατύπωση. Βεβαίω ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιες οδοί που έχουν σημαντική κίνηση και έχουν αναπτυχθεί, Άλλε όμω θα πρέπει να βελτιωθούν και να διευρυθούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η προθεσμία είναι 27 Ιουλίου στις 12 για τις ε, τροπολογίες. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάτεξης, την Ευρωπαϊκή Στρατηγική ε, για το φυσικό αέριο, το υγροποιημένο φυσικό αέριο και την αποθήκευση φυσικού αερίου. Η Κλαούντιο Μοντέιρο Ντεμουιάρ είναι η συγγήτρια και έχει το λόγο. Ε, Sr. Presidente. Eh, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, σε σχέση με την έκθεση αυτή, να αναφέρω δύο παρατηρήσεις. Καταρχάς, θα ήθελα να αναφερθώ στο ζήτημα της ενεργειακής αυτονομία της Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω πως χρειαζόμαστε μια αγορά η οποία θα είναι πιο διαφανής ε, και μια ε, αγορά η οποία ε, προάγει λιγότερο τις διακρίσεις. Θα πρέπει να έχουμε μια καλύτερα, μεγαλύτερη ικανότητα των σχετικών σταθμών ανεφοδιασμού και στους ευρωπαϊκούς λιμένους και θα πρέπει βέβαια να αυξήσουμε τη σημασία των ε, περιφερειακών ε, λιμένων και να προωθήσουμε περισσότερο τη συνδεσιμότητα. Νομίζω πως ε, το υγροποιημένο φυσικό αερό μπορεί να αποτελεί μια ευκαιρία για να μειώσουμε τις εκπομπές του άνθρακα στην οικονομία μας και τη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου έχουν υποβληθεί 23 τοπολογίε για τη συγκεκριμένη έκθεση και και έχουμε ε, συμβαστικές τροπολογίες οι οποίες έχουν υιοθετηθεί από το σύνολο όσων συμμετείχαν. Άρα λοιπόν πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας ε, κοινή εργασίας σε αυτό το κείμενο και γιατί πραγματικά με την πολύ καλή συνεργασία είχαμε την ε, συμβολή από την πλευρά των συναδέλφων έτσι ώστε να έχουμε μια ένα ενιαίο ρόμα σε ό,τι αφορά το ρόλο ε, του υγροποιημένου φυσικού αερίου στον τομέα ε, τις οικονομίες, χωρίς βέβαια να ξεχνάμε τις περιβαλλοντικές ε, πτυχές ε, και γίνεται και εδώ και μία αναφορά στην χρηματοδότηση την οποία θεωρούμε απαραίτητη. Επιτρέψτε μου να αναφέρω για μία ακόμα φορά το γεγονός ότι τονίζουμε εδώ τον κρίσιμο ρόλο που θα κληθούν να παίξουν οι λιμένε. Ε, δηλαδή, είναι ε, απαραίτητοι οι λιμένε προφανώ για τη ε, φόρτωση εισαγωγή και εξαγωγή, αλλά και ακριβώ για τον ανεφοδιασμό των πλοίων με το ντροπημένο φυσικό αέριο. Επίση, αναφερόμαστε για μία ακόμα φορά στην ανάγκη σωστή εφαρμογή τη οδηγία σε ό,τι αφορά τα εναλλακτικά καύσιμα και έω τι 18 Νοεμβρίου θα έχουμε τη δυνατότητα για την υποβολή των υπολογιών. Και εκείνο που αποτελεί το την απόλυτη προτεραιότητά μα είναι η βελτίωση των συστημάτων αποθήκευση και μεταφορά του υγροποιημένου φυσικού αερίου χωρί να ξεχνάμε τις παραγωγικέ πτυχέ, και όπω ε, ε, είπα ήδη θα πρέπει να επιμείνουμε στη σωστή εφαρμογή τη οδηγία για τα εναλλακτικά καύσιμα. Θα πρέπει προφανώ ε, να προωθήσουμε και τι ε, κλίμακες επενδύσει επενδύσεις σε υποδομές να προωθήσουμε τη συνδεσιμότητα για παράδειγμα και μέσω τη νησού και όποια άλλα εργαλεία έχουμε στη διάθεσή μας από εκεί και μετά. Ε, ναι, ε, σας υπενθυμίζω την πρόταση που κάναμε σε ό,τι αφορά τα, τη χρήση των blue corridors για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, σε ό,τι αφορά τις απομακρυσμένες ε, περιοχές και τις νοσητικές περιοχές και τη σύνδεσή τους με τις ε, ε, υπηρετικές Θα πρέπει να προωθήσουμε την κατασκευή των ε, σταθμών ανεφοδιασμού ε, και ε, μεταφοράς και θα πρέπει να δημιουργήσουμε και να διασφαλίσουμε τα κατάλληλα ε, κίνητρα ε, για την χρήση αυτής της τεχνολογίας μέσω του retrofitting, δηλαδή της εκ των κατάστασης του, σχετικού εξοπλισμού. Αλλά για να επιτευχθούν όλα αυτά θα πρέπει προφανώς ε, τα project κοινού ενδιαφέρον στον ενεργειακό τομέα να λάβουν την κατάλληλη υποστήριξη των κρατών μελών και να δοθεί και κατάλληλη πρόσβαση στην αγορά. Νομίζω πως ένα σημαντικό στοιχείο είναι να υπάρχει η, ακριβώς η δυνατότητα εμ, ροής, αμφίδρομης ροής ε, του αερίου μεταξύ των χωρών, τόσο ώστε να έχουμε καλύτερη διανομή. Νομίζω πω με αυτόν τον ε, τρόπο μπορούμε να προωθήσουμε καλύτερο το θεματολόγιο, το μίξ, το ενεργειακό μίξ που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε ένα ενιαίο σύστημα με την κατάλληλη χρηματοδότηση ε, και αξιοποιώντα ε, ταυτόχρονα τις δυνατότητες που, που έχει ήδη ο Διεθνή Αυτολιστικός Οργανισμό και η δική μα Ευρωπαϊκή Αρχή σε αυτό το τομέα. Νομίζω πως ε, ε, με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να επιτύχουμε έναν ε, κοινό στόχο, δηλαδή να έχουμε μια στρατηγική η οποία θα είναι πιο ευέλικτη, θα επιτρέπει δηλαδή περισσότερε αναλλακτικέ λύσει και θα, έχει, θα είναι πιο συμμετοχική για όλου. Ευχαριστώ. Η συγκήτριά μα είναι από την Πορτογαλία και βλέπω πω η ένδυσή τη αποτελεί μια ένδειξη σε ό,τι αφορά την, την νίκη τη Πορτογαλία στο πρωτάθλημα, οπότε τα συγχαρητήριά μα. νομίζω πω είναι πρώτη φορά ε, που παίρνει το πρωτάθλημα και μάλιστα στο 65ο λεπτό χωρίς τον Ρονάντο. Ποιος θα το περίμενε. Ε, Τζάκι Φώστερ έχει τώρα το λόγο. I wouldn't Τα καταφέρατε, μπράβο. Ε, ναι, συγχαρητήρια. Συγγνώμη, Τζάκι, μισό λεπτό. Ρεβόντα πρώτα. Όχι εγώ, μάλιστα. Oui, euh... Η Τερέζα δεν μπορεί να έρθει και μου ζήτησε να την συγχωρήσετε και θα ήθελα καταρχάς να πω επειδή ήταν πολύ καλό το μάτς ε, χθες, ε, να ευχαριστήσω, να πω μπράβο σε αυτή την πολύ καλή ομάδα της Πορτογαλίας. Θα το πω γιατί υποστήριζα τη Γαλλία μέχρι τέλους, αλλά ήταν πολύ καλή ομάδα σας. Να πω λοιπόν αυτό που ήθελε να πει η Τερέζα. Καταρχάς ήθελε να ευχαριστήσει την, Κλόντια για την, πολύ, την Κλαούντια για την πολύ καλή δουλειά που έκανε ω τώρα και τις συμβαστικές τροπολογίες. Χαίρεται για την ε, αναφορά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αφαίρεση του άνθρακα από την οικονομία των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Θεωρεί ότι πρέπει να φτιάξουμε μια στεναρή ένωση για την ενέργεια και το υγροποιημένο φυσικό αέριο να βοηθήσει στη βιωσιμότητα αυτής της αγοράς. Στην ομάδα των σκιωδών τέθηκαν κάποιες προτεραιότητες που έλαβε υπόψη της εισηγήτριας συγκεκριμένα να είμαστε ε, σόφρονος ως προς την ανάπτυξη των υποδομών, ε, οι νέες υποδομές δηλαδή να αντικατοπτρίζουν την πραγματική ζήτηση σε αέριο. Επίσης ε, θα πρέπει να γίνει πιο σωστή χρήση των σταθμών που υφίστανται ήδη για το ευρωποιημένο φυσικό αέριο. Η ομάδα μας, για να καταλήξω, θεωρεί ότι πρέπει να θυμίσουμε στην Κομισιόν τις συνεχείς εκκλήσεις του ε, Κοινοβουλίου για, τις φιλόδοξες, ε, για τους φιλόδοξους στόχους, τους περιβαλλοντικούς ε, για το 2030. Ευχαριστούμε την Κλόντι για την πολύ καλή ε, εισήγησή της. Ευχαριστούμε και τώρα η Τζάκη Φώστερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την εισηγήτρια. Θα πω μόνο λίγα πράγματα σχετικά με την Συμβαστική 1. Νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ συμφωνούν με τον τρόπο που θα προχωρήσουμε. Πρέπει να βρούμε εναλλακτικέ και ο θαλάσσιος τομέας είναι πολύ σημαντικός γι' αυτό όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ανανεώσιμες και πιο καθαρά καύσιμα, θα το κάνουμε και πρέπει να το θέσουμε αυτό το θέμα. Επίσης έχω μια μικρή ανησυχία σε σχέση με δύο-τρεις συμβαστικές λύσεις. Μία από αυτές φαίνεται να πηγαίνει πέρα από αυτά που λέει η οδηγία για, τις για τα εναλλακτικά καύσιμα. Μας ανησυχεί λίγο αυτό γιατί υπάρχει οδηγία για τα εναλλακτικά καύσιμα ήδη. Άρα, αν αρχίσουμε να βγαίνουμε εκτός του πεδίου του θέματος δηλαδή που εμείς πρέπει με το οποίο πρέπει να ασχοληθούμε σε κάθε περίπτωση θα είναι δύσκολο και κακό. Θυμάμαι στο παρελθόν που είχαμε μια παρόμοια συζήτηση για μια παρόμοια έκθεση στην οποία εγώ έλεγα ότι τα ίδια τα κρατημέλη έπρεπε να ορίζουν τα, τα καύσιμα που θέλουν και τις απαιτήσει τους και να μην είμαστε τόσο εμείς ε, ε, ρυθμιστικοί. Και νομίζω ότι τελικά καταφέρουν τα κράτη-μέλη να κάνουν ε, αυτό που έπρεπε και πρέπει να αφήσουμε την αγορά να προχωρήσει ελεύθερα. Τώρα για τις περιβαλλοντικές λύσεις θεωρώ ότι και πάλι πρέπει να έχουμε παρόμοια κριτήρια. Πάλι η αγορά πρέπει να λύσει το ζήτημα. Αυτό ήταν ε, η συμβαστική μας προσέγγιση τόσο ή άλλως. Χαίρομαι ότι ε, και από την ε, πλευρά της Επιτροπής Ιντρα θα μπορέσουμε να έχουμε μια καλή κατάληξη ως προς την γνωμοδότηση που θα δώσουμε. Ευχαριστώ. Ιούζο Ράντος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο βασικός ε, στόχος ε, της στρατηγικής για το υγροποιημένο φυσικό αέριο είναι ξεκάθαρος. Μπορεί να πραγματοποιηθεί, θεωρώ. Πολλές ομάδες έχουν καταθέσει διαφορετικές τροπολογίες ε, σχετικά με την χρήση στον τομέα των μεταφορών και Έχουμε μεγάλο πεδίο, έχουμε τη μαζική χρήση του LNG. Εγώ το υποστηρίζω το θέμα αυτό, όμως παραμένει ένα ζήτημα ανοιχτό. Ποιο είναι το αέριο. Το, έχουμε το υγροποιημένο, αυτό που είναι υποποίηση, αυτό που γίνεται μέσω απόσταξης ή βιοκαύσιμα. θε τίθεται λοιπόν το ερώτημα ποια είναι η βέλτιστη λύση, ποιο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Επίσης πρέπει να δούμε αν όλα αυτά είναι συμβατά, αν υπάρχουν ήδη νέες τεχνολογικές λύσεις. Όπως και να έχει, η ομάδα ALDE υποστηρίζει το μεγαλύτερο κομμάτι των κατατεθισών τροπολογιών, όμως για μένα παραμένει το ερώτημα του πώς θα αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι θα υπάρχει μαζική χρήση του LNG στον τομέα των μεταφορών. Ευχαριστώ. Ο επόμενο ομιλητή ο Keith Taylor. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ζητώ συγγνώμη που άργησα λίγο. Αρχίσατε λίγο νωρίτερα από ό,τι έλεγε το πρόγραμμα, αλλά όπως και να έχει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τους σκιώδεις και την καλή συνεργασία σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν κάποιες ε, καλές προσεγγίσεις σε αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης. Καταρχάς το γεγονός ότι το LNG δεν πρέπει να πάρει τη θέση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ότι πρέπει η παραγωγή να είναι αϊφόρος, βιώσιμη και να ε, συνεισφέρει στη μείωση των εκπομπών διεξιδίου του άνθρακα. Επίσης χαίρομαι για την αναγνώριση του γεγονότος ότι η στρατηγική για το LNG πρέπει να ταιριάζει με την COP21 και τη γενικότερη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα περιβαλλοντικά, για τη μείωση της ζήτησης, για την απο... αποτελεσματική... αποτελεσματική ενέργεια και για τα ορυκτά καύσιμα και τη μείωση της χρήσης τους μέχρι το 2050. Επίσης, να πω ότι παρόλα αυτά μιλάμε για το LNG με ενθουσιασμό σαν μια βιώσιμη λύση για την αντικατάσταση των παραδοσιακών καυσίμων. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το LNG έχει λιγότερη, ε, λιγότερες εκπομπές σε διοξείδιο του άνθρακα, σε θείο, σε άζωτο από ότι τα παραδοσιακά καύσιμα, όμως παραμένει ορυκτό καύσιμο πρέπει αυτό να χρησιμοποιηθεί ως μεταβατικό εργαλείο και πρέπει να το τονίσουμε. Επίσης πρέπει να είμαστε αναλογικοί σε σχέση με τα ε, ωφέλη που μπορούμε να έχουμε στον τομέα των μεταφορών από την χρήση του LNG. Το σχέδιο της γνωμοδότησης επίσης κατευθύνεται προς την παροχή κινήτρων προς την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη για να ε, δημιουργήσουν περισσότερες υποδομές LNG που εγώ θεωρώ ότι είναι μεγάλο η ανησυχία. Το ίδιο κάνουν και οι τροπολογίες. Επίσης θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι το φυσικό αέριο δεν μπορεί να μας βοηθήσει να μειώσουμε τις εκπομπές διεξιδίου του άνθρακα στο βαθμό που θέλουμε στις μεταφορές για να φτάσουμε στους στόχους που έχουμε θέσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέχρι το 2050. Έχουμε περιορισμένα ωφέλη και υπάρχει κίνδυνος η επένδυση, οι περισσότερες επενδύσεις σε LNG να μας κάνει να παρεκτραπούμε από τις πραγματικές εναλλακτικέ με χαμηλές επενδύσεις, ε, με χαμηλές εκπομπές και να έχουμε υπερεπενδύσεις που θα μας φέρουν σε διέξοδο. Επίσης υπάρχει μια ουδετερότητα της τεχνολογίας που πρέπει να χρησιμοποιηθεί και αυτό φαίνεται ότι δεν θίγεται πρέπει να έχουμε περισσότερες επενδύσεις δημοσίων πόρων ε, για τη βιώσιμη ηλεκτροδότηση και ε, για τις βιώσιμες λύσεις ε, που θα είναι πραγματικά εναλλακτικές πηγές ενέργειας, ανανεώσιμες. Επίσης, το σχεστολιστικό αέριο είναι μία από τις πιθανότητες για την παραγωγή σε αυτήν εδώ την περίπτωση και αυτό με ανησυχεί ιδιαίτερα. Να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια λοιπόν άλλη μια φορά και τον πρόεδρο. Και έχετε το λόγο. το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ την Κλάουδα για τις εξαιρετικές ε, συμβαστικές τροπολογίες που μας έχει ε, προτείνει και ε, οι οποίε με καλύπτουν σε ό,τι αφορά τι δικέ μου τροπολογίε. Θα ήθελα να επισέλθω σε κάποια ζητήματα. Σε ό,τι αφορά τα εναλλακτικά καύσιμα γενικά, η χρήση του ε, πάντοτε εξαρτάται από τη χρήση και τη κατάλληλη υποδομή η οποία δεν προβαίνει σε διακρίσει ό,τι αφορά του χρήστου. Η πολυτροπικότητα των σχετικών του, του αερίου είναι ιδιαίτερη ιδιαίτερα χρήσιμη γιατί ακριβώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να μεταφερθεί με διάφορα ε, οχήματα και μέσω τη ναυσιπλοεία και ε, βαρέου τύπου και ούτω καθεξή. Νομίζω λοιπόν πω θα πρέπει να επενδύσουμε σε όλου του ε, τρόπου μεταφορών και μεταξύ αυτών και μεταφορά του LNG και εκείνο που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι η σιδηροδρομική μεταφορά του υγροποιημένου φυσικού αερίου γιατί με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσαμε περισσότερο καύσιμο και μάλιστα τη μεταφορά του με βιώσιμο τρόπο ακριβώ, δηλαδή μέσω σιδηροδρομικών μεταφορών ε, εγώ ε, ευχαριστώ λοιπόν την εισηγήτρια, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τι συμβαστικέ τροπολογίε και την ε, αποδοχή τη τροπολογία 90 από δική μου πλευρά. Ε, κυρία Ζαμπέλα, δεν μου το έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Καταρχά, διπλά συγχαρητήρια στην εισηγήτρια και για το ποδόσφαιρο και τα αποτελέσματα, αλλά και για το αποτέλεσμα τη νομοδότηση. Νομίζω ότι είναι για μένα σημαντικό να υπάρχει παρόμοια προσέγγιση, γιατί αυτό καταδεικνύει ότι δεν αντικαθιστούμε τις ανανεώσιμες, αλλά αναγνωρίζουμε ταυτόχρονα τη σημασία των αλλακτικών καυσίμων όπως αυτό εδώ. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόσφατα, όταν αξιολογήσαμε το REFIT σε σχέση με τα σχέδια συλλογής των πλοίων, των απορριμμάτων των πλοίων, αναγνωρίσαμε ότι τα αποτελέσματα της οδηγίας δεν ήταν βελτιστά δεν ήταν τα καλύτερα δυνατά. Οπότε η επένδυση σε εναλλακτικά καύσιμα και σε πιο βιώσιμα καύσιμα είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης θεωρώ ότι είναι ουσιώδες να υπάρχει ανεφοδιασμός όχι μόνο στα λιμάνια αλλά και σε διάμεσους λιμένες μέχρι να υπάρχει πλήρης πρόσβαση. Αλλά για να γίνει αυτό θα είναι πολύ δύσκολο όποιος διαθέτει ένα όχημα, όποιος έχει ας πούμε ένα φορτηγό να κάνει μια πλήρη μετατροπή του στόλου του. Οπότε είναι σημαντικό να υπάρχει πλήρης διάθεση, διαθεσιμότητα. Και είναι απαραίτητο να υπάρχει βέβαια και ένα σταθερό χρηματοδοτικό πλαίσιο. Εγώ συμμετείχα στις εκδηλώσεις του 20 Days. Εκεί οι ενδιαφερομένοι μας μίλησαν για τις επενδύσεις και μας παραπονέθηκαν για το ότι δεν έχει δοθεί ακόμα διέξοδο στις επενδύσεις τους. Θα πρέπει λοιπόν μεταξύ των διαφόρων κονδυλίων των ταμείων να γίνεται για μια σύγκριση όσον αφορά τα καύσιμα. Επίσης, να πω για τις τροπολογίες, για την 8 συγκεκριμένα, όπου μιλάμε για τη γεωργία. Εκεί έχουμε κάνει βήματα προόδου όσον αφορά τη μείωση των τρύπων. Και μετά για τις 48 να πω εκεί που ζητάμε δηλαδή την ε, βελτιστοποίηση, την διασυνορική αυτονομία, χωρίς να έχουμε νέες μονάδες υγροποίησης του αερίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ πρόεδρε. ξέρω ότι σήμερα δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους οικειοδησίκτες γιατί πραγματικά ήταν ε, πολύ καλέ οι προτάσει, δηλαδή και στην Ήτρε ε, και στην Envy ε, και εδώ συζητάμε σήμερα το LNG, δηλαδή είναι η μέρα του LNG πραγματικά. αυτό που υπόθηκε είναι πολύ σωστό, δεν αποτελεί πανάκια, αλλά αποτελεί μια πρόοδο όταν έχουμε να κάνουμε με μείωση των εκπομπών. Και αυτό το διαπιστώσαμε ειδικότερα ε, στον τομέα της ναυσιπλοείας, δηλαδή στα καράβια τα οποία χρησιμοποιούν για παράδειγμα στην ε, ε, Βαλτική αυτή την περίοδο LNG και πώς μειώθηκαν εκεί οι εκπομπές. Έχουμε ακριβώς αποφασίσει μια πολιτική για τις εναλλακτικέ πηγές ενέργειας και πράγματι αυτά τα εναλλακτικά καύσιμα μπορούν να μεταφερθούν και με τους σιδηροδρόμους και με πλοία και ακριβώς το ζήτημα σε σχέση με την ανάπτυξη των υποδομών είναι και η να έχουμε χρήση ε, πλοίων ε, και βέβαια ε, έχουμε αυτή την ευελικτία. Δηλαδή, με την παρότι δεν πρόκειται για πανάκια, θα πρέπει ε, να δούμε ότι να, διαπιστώσουμε ότι πραγματικά έχουμε τι ε, απαραίτητε υποδομέ και θα πρέπει από εκεί και μετά, με βάση βέβαια το όσο έχουμε προβλέψει, να δούμε κατά πόσο έχουμε αξιοποιήσει αυτή την υποδομή. Δηλαδή να μην οδηγηθούμε σε μια κατάσταση όπω έχει γίνει και στη Γερμανία, όπου λέμε ότι δεν υπάρχει η υποδομή ε, για να εφαρμόσουμε αυτή την τεχνολογία. Θα πρέπει αυτή την περίοδο που βρισκόμαστε σε τόση ευρωδημασία να ε, διασφαλίσουμε την επίτευξη των ε, στόχων μας. Ε, και προφανώς ε, το καλύτερο θα ήταν να έχουμε βιοκαύσιμα για να επιτύχουμε και τους στόχους από την COP21 και όχι υγροποιημένο φυσικό Αλλά από την άλλη πλευρά το βιοκαύσιμο αποτελεί κατά κάποιο τρόπο βέβαια ένα υποπροϊόν μέσα της διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση όμως η αποτελεί μια βιώσιμη εναλλακτική λύση ε, το ε, υγροποιημένο φυσικό αέριο και θα πρέπει να το χρηματοδοτήσουμε χωρίς όμως να αποτελέσει τη λύση για τα πάντα. Ε, ευχαριστώ. Θα μιλήσω εξ ονοματός μου. Ναι, νομίζω ότι εδώ μπορούμε να μιλήσουμε για εναλλακτικά καύσιμα. σε σχέση με τους στόχους του περιβαλλοντικού και τη λευκή βίβλο για τις μεταφορέ. Είναι σημαντικό λοιπόν η Κομισιόν μα να θετήσει ένα φιλόδοξο στόχο για το αέριο. Πολλά θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε εδώ και να κάνουμε. Καταρχάς, να μιλήσουμε για το υγροποιημένο που προέρχεται από τις... το αέριο προέρχεται από τις ανανεώσιμες. Μετά θα πρέπει να μιλήσουμε για την αναθεώρηση των οδηγιών που αφορούν τις ΑΠΕ και την ποιότητα των καυσίμων, ώστε να κάνουμε συγκεκριμένες δημοθετικές συστάσεις για την αύξηση των βιοκαυσίμων και του αερίου, ζητώντα από την Κομισιόν βεβαίω καταρχά να θεσπίσει στόχου για μετά το 2020 όσον αφορά τι ΑΠΕ στι μεταφορέ μέχρι το 2030 και να έχουμε και ένα νέο στόχο μετά το 2020 σε σχέση με την μείωση του άνθρακα στις μεταφορές. Αυτές λοιπόν οι συγκεκριμένες συστάσεις θα έπρεπε να περιλαμβάνουν και την αναφορά στην ανάγκη υλοποίηση ενός αντιστοίχου διοξιδίου άνθρακα, δίκτυ διεξιδίου άνθρακα για τα βιοκαύσιμα που θα χαροποιήσει του κατανάλωτε Ελπίζω αυτέ τις προτάσεις μου να βρουν θέση στην τελική μορφή του γράφου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, Παίρνω τελευταίο ε, το λόγο και να πω και εγώ ε, ότι ναι και είναι να έχει δίκιο. Δηλαδή χρειαζόμαστε όλε τι αναλλακτικέ. Το ευρωπημένο φυσικό αέριο ε, δεν αποτελεί πανάκια, αλλά πραγματικά υπάρχει, πρόκειται για ένα κάψιμο το οποίο δεν απαιτεί την αλλαγή τη υποδομή. Αλλά πραγματικά αποτελεί ε, ε, μια καλύτερη ανακριτική σε σχέση με το βαρύ πετρέλαιο, το οποίο βαρύ πετρέλαιο ε, πραγματικά αποτελεί προϊόν και το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο σε σύγκριση με το φυσικό αέριο. Ειδικότερα δηλαδή και το ντίζελ δεν αποτελεί κάτι το θαυματουργό, αλλά εάν συγκρίνουμε το ντίζελ με το βαρύ πετρέλαιο, θα δούμε το αργό πετρέλαιο, δηλαδή θα δούμε ότι πραγματικά είναι καταπληκτικό το ντίζελ. Τι σημαίνει και για, το, και για αυτή την περίπτωση για το φυσικό αέριο, θα πρέπει να έχουμε ε, την αξιοποίηση της υποδομής που ήδη έχουμε στα χέρια μας, αλλά από εκεί και μετά θα πρέπει να έχουμε την απόρριψη με βάση τον τρόπο που προβλέπετε Δηλαδή θα πρέπει ε, να έχουμε την κατάλληλη χρηματοδότηση χωρίς να πάρουμε τα κονδύλια από αλλού και να πούμε ότι ε, να απαγορεύσουμε το, το, το, ταχύτερο δυνατό, το ταχύτερο δυνατό γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε τόσο γρήγορα, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας γιατί ούτως ή άλλως οι εκπομπές σε παγκόσμιο επίπεδο αφορούν και εμάς και στο ίδιο πλαίσιο θα πρέπει να δούμε τις εναλλακτικέ που έχουμε στη διάθεσή μα μεταξύ αυτών και το φυσικό αέριο. Ε, ο λόγο ε, τώρα στον Αντώνιο Τρίκα από τη Γενική Διεύθυνση ΜΟΥΚ τη Επιτροπή. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ λοιπόν για τις τροπολογίες σας. Συμφωνούμε με το περιεχόμενο αυτό των τροπολογιών και συμφωνούμε με τα περισσότερα σχόλια που ανέφεραν τα αξιότυπα μέλη της Επιτροπής. Θεωρούμε ότι το ευρωποιημένο μπορεί να βοηθήσει συγκεκριμένες μορφές μεταφορών, θαλάσσιες, βαριές μεταφορές κλπ. Επίσης, συμβάλλει στη μείωση ρήπων όταν αναμεγνύεται με βιομεθάνιο ή συνθετικό φυσικό αέριο από ανανεώσιμες. Επίσης θεωρούμε ότι το LNG παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα στη μείωση ρήπων όπως θείο, άζωτο κλπ. που συναντούνται ιδιαίτερα στον θαλάσσιο τομέα, στις θαλάσσιες μεταφορές σε σημαντικό ποσοστό, 30 αντίστοιχα. Θέλει να προωθήσει το LNG η και αυτή τη στιγμή δουλεύουμε πάνω στην εφαρμογή της ε, οδηγίας. Οι χώρες μέλη πρέπει να υποβάλουν μέχρι τον Νοέμβρη φέτος το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο και επίσης ε, εργαζόμαστε πάνω σε πρότυπα και η ΕΜΣΑ κάνει το ίδιο με την εκπόνηση εγγράφων κατευθυντήριων γραμμών για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Έχουμε και ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, τη διευκόλυνση, που προβλέπει τις υποδομές ε, LNG όσον αφορά κυρίως τις θαλάσσιες μεταφορές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο εισηγητής για άλλη μια φορά. Παρακαλώ. Ε, Πρωταθλήτη Ευρώπη στη Σίγητρα έχει Ευχαριστώ. Και σας ευχαριστώ και για τα συγχαρητήριά σας ε, για, τον, ε, για την ομάδα μας και παρότι δεν ε, ήταν ε, εκείνη την ώρα μέσα στο γήπεδο Ρονάντο, ε, μας βοήθησε και εκτός γήπεδου να κερδίσουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ε, συναδέλφους που ε, μας, ε, με βοήθησαν στο πλαίσιο της προετοιμασίας αυτής της γνωμοδότησης και προφανώς θα λαφθούν υπόψη τα εν λόγω σχόλια. Ε, αλλά πραγματικά πρόκειται εδώ για μια γνωμοδότηση η οποία είναι συνενετική και η οποία παρουσιάζει ακριβώς μια στρατηγική ε, ως προς την αξιοποίηση των διαφορετικών εναλλακτικών που έχουμε ε, για την αξιοποίηση των ενεργειακών μας ε, πηγών. Άρα λοιπόν θα, λάβουμε, θα λάβω υπόψη τα σχόλια και ευχαριστώ για μία ακόμα φορά για τη συμβολή των συναδέλφων και βέβαια και τη γραμματεία γιατί πραγματικά η βοήθειά της ήταν κεντρική σημασία για να επιτύχουμε την προετοιμασία αυτή. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. 5η 1η Σεπτεμβρίου είναι η προθεσμία όπου θα έχουμε δηλαδή την ψηφοφορία. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημέρας διάταξης που είναι οι τεχνικές προδιαγραφές για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοείας, ο λόγος των Ιβο Μπέλετ. Ευχαριστώ, ε, Μάικλ. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω περί τίνος ε, πρόκειται ε, και από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, οπότε θα είμαι πολύ σύντομος. Νομίζω πως στην, στο σημείο 9 και ειδικότερα στην ετελογική εκεί έκθεση μπορείτε να δείτε τι ακριβώς κάναμε μέσα στο τελευταίο χρόνο σε ό,τι αφορά την εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοείας. Πρόκειται για μια διαδικασία που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια με την Karen Corpan Calls με μια πρώτη έκθεση όπου είχαμε σκεφτεί ότι α, θα είναι πολύ εύκολο και θα τελειώσουμε μέσα σε λίγους μήνους αλλά τελικά ξεκίνησε εκεί μια η ε, υπηρεσιακή, αν θέλετε, μια ε, διαθεσμική ε, διαμάχη, να μην την πω διαμάχη, αλλά πάση περιπτώσει μια μακρά συζήτηση με το Συμβούλιο και τελικά φτάσαμε σε ένα αρκετά ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Έγιναν διαπραγματεύσει υπό την Προεδρία του Λουξεμβούργου και των κάτω χωρών. Πραγματικά υπήρξε μια πάρα πολύ κοινή συνεργασία, ειδικότερα με την Ολλανδική Προεδρία και την οποία θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω για την επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεων. Το πιο σημαντικό ζήτημα ήταν βέβαια το θέμα των της πράξεων. Όπως γνωρίζετε, ε, το εν λόγω ζήτημα αποτέλεσε το πρώτο σημείο στο πλαίσιο του οποίου εξετάστηκε ακριβώς αυτή η δυνατότητα ε, των κατεξοδότηση πράξεων στο πλαίσιο της Συμφωνία. Ε, ε, συμφωνίας. Εδώ λοιπόν για πρώτη φορά τέθηκε σε δοκιμή αυτή η νέα συμφωνία και όταν είχε πριν από 1,5 χρόνο προς προταθεί από το Συμβούλιο να υπάρχει μια δυναμική αναφορά σε ό,τι αφορά στην ενημέρωση των τεχνικών του προδιαγραφών, υπήρχε μια, μια αμφιβολία από την πλευρά ε, του Συμβουλίου γιατί θεωρούσε ότι το Συμβούλιο, ότι το Κοινοβούλιο θα παρεμβαίνει ξανά και ξανά ε, στο πλαίσιο των ενημερώσεων που θα γίνονται. Εμείς γι' αυτό το λόγο ε, προτείναμε και αυτή την εναλλακτική. Το Συμβούλιο επίσης είχε προτείνει και μία ρήτρα διασφάλιση, ένα safe cut clause, με βάση το οποίο όπου δεν υπάρχουν πρότυπα περιβαλλοντικού χαρακτήρα ή όπου υπήρχε κίνδυνο για την ασφάλεια. Αυτό ε, αρχικά θεωρήθηκε πω αποτελεί μια καλή λύση, αλλά μετά διαπιστώθηκε ότι δεν θα υπήρχε λόγο να ε, ενεργοποιηθεί αυτή η safeguard clause και κατά συνέπεια δεν μπορούσαμε να την κάνουμε δεκτή γιατί δεν θα μπορούσε να συμπεριληφθεί μέσα στη διαδικασία λήψη των αποφάσεων. Ε, διαπραγματευτήκαμε λοιπόν με το Συμβούλιο και φτάσαμε σε αυτή τη λύση που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας, δηλαδή να επιλέξουμε τις και της πράξη. Νομίζω πως με αυτό το αποτέλεσμα λοιπόν του τριμερούς ε, διαλόγου θα έχουμε την εφαρμογή αυτών των εποσμανόμενων ε, προτύπων της ΣΕΣΜΗ. Και νομίζω ή μάλλον όλες οι ε, αλλαγές από εδώ και στο εξή θα λαμβάνουν χώρα το τεχνικό μετεωρό θα λαμβάνουν χώρα μέσω τη κατεξοδότηση πράξη. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίσαμε τρία πράγματα. Πρώτον, ότι θα υπάρχουν εναρμονισμένα πρότυπα σε αυτό το τομέα που αποτέλεσε βέβαια και το βασικό στόχο αυτή τη ε, νομοθετική ε, πρωτοβουλία. Ύπαρξη λοιπόν εναρμονισμένων ε, προτύπων σε όλα τα κράτη-μέλη και στις οδούς εσωτερικής να σε όλα τα κράτη-μέλη. Δεύτερο στοιχείο είναι ότι αποφεύγουμε περαιτέρω διοικητικό άκτο, το οποίο αποτέλεσε βέβαια και ε, μία από τι ε, θεμητέ ανησυχίε του κλάδου, που δεν ήθελαν δηλαδή να δημιουργηθεί ακόμα περισσότερη γραφειοκρατία. Έτσι λοιπόν επιτύχαμε ακριβώ αυτό, να μην υπάρξει επιπρόσθετο διοικητικό άκτο και τρίτον, καταφέραμε να διασφαλίσουμε όλες ε, τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο ακέραιο. Οπότε θα ήθελα να καλέσω ε, την Επιτροπή μας να να γνωρίσει την πρώτη ανάγνωση εδώ, την οκλήρωση τη πρώτη ανάγνωση ε, του Συμβουλίου και να συμφωνήσει με τι προτάσει που κάνουμε εμεί από την πλευρά μα στο πλαίσιο τη δεύτερη ανάγνωση προ το Συμβούλιο. Μάικλ, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω εμφατικά γιατί έπαιξε πολύ κεντρικό ρόλο στο πλαίσιο αυτή τη διαδικασία. Σε ευχαριστώ λοιπόν και ευχαριστώ όλου του συντονιστέ, ε, ευχαριστώ όλου του συναδέλφου και τι συζητητέ που συμμετείχαν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την γραμματεία τη ε, Επιτροπή ΕΤΡΑΝ, ειδικότερα τον Ντομινίκ Ντομινίκ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, για το εξαιρετικό έργο που έκανε μαζί με την νομική υπηρεσία. Ευχαριστώ όλου του συμβούλου όλων των πολιτικών ομάδων, ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, την ε, Ολλανδική Προεδρία για αυτή την πραγματικά εξαιρετική δουλειά που κάναμε. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου εγκάρδια ε, στο όλο σου γιατί χωρί εσένα δεν θα είχαν πάει πολύ καλά τα πράγματα. Πραγματικά ήταν πολύ καλή η συνεργασία μα και τα καταφέραμε ε, να επιτύχουμε αυτά που θέλαμε και ε, ήταν πολύ καλό το αποτέλεσμα. Δεν είχε προβλεφθεί συζήτηση για αυτό το σημείο, αλλά αν υπάρχουν κάποια επίγοντα σχόλια από κάποιου συνάδελφου, μπορεί να τα κάνει. Ο παρακαλώ. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή για θαυμάσια δουλειά του και κυρίως για τις προσπάθειες διασφάλισης των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου ως συνομοθέτη. Αυτά και για τις ε, τροπολογίες επίσης, ε, για την προθεσμία. Ευχαριστώ η Γεζίνε. Ήταν πολύ δύσκολη αυτή η νομοθετική πράξη και ήταν δύσκολο να επρασπιστούμε τα δικαιώματά μας. Ε, τα καταφέραμε πολύ γιατί είχαμε πολλούς διπλωμάτες και η Ολλανδία βοήθησε πάρα πολύ. Ήταν καλό και χαίρομαι που λειτουργήσε έτσι, αλλιώ δεν θα μπορούσαμε να καταφέρουμε αυτό που θέλουμε. Ευχαριστώ, λάμπω μου από χαρά. Να πω κάτι που πρέπει ως πρόεδρος. 14 Ιουλίου είναι η ημερομηνία για τις τροπολογίες στις 12 η ώρα. Όμως, να πω ότι αυτή η αλλαγή ημερομηνία στην ουσία είναι τυπική γιατί ήδη υπάρχουν τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου. Οι τροπολογίες μπορούν θεωρητικά να κατατεθούν στη δεύτερη ανάγνωση, όμως ε, θα κατέστρεφαν το συμβιβασμό ε, ακόμα και αν ε, γινόταν αποδεκτή και μία τροπολογία. Υπάρχει λοιπόν δυνατότητα για τις τροπολογίες, αλλά πρέπει να ξέρουμε τις επιπτώσεις. Ήδη ως πρόεδρος έχω ενημερώσει το Συμβούλιο για την ψηφοφορία μας, να το ξέρετε, το ξέρει. Αυτό απλώς προς πληροφόρησή σας. Έχουμε το δικαίωμα, ελπίζω να μην ε, υπάρξουν όμως τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ωραία, πάμε τώρα την ε, πρόσβαση ε, στις, στα, στους λιμένες είναι μια έκθεση του κυρίου Φλεκενστάιν που δεν είναι εδώ. Α, εδώ είναι. Κνούτ, δεν σε είχα Ζητώ συγγνώμη, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ. Θα πω δύο πράγματα. Στη είχαμε στις 24 του Ιουνίου ε, πετύχει μία, ένα συμβιβασμό με την Ολλανδική Προεδρία. Βέβαια δεν τα καταφέραμε όλα, αλλά τα περισσότερα. Γι' αυτό έχουμε την ανάγκη ε, να ευχαριστήσουμε τους συγκητές από το ΕΛΚ, το ΑΛΤΕ, τους Πρασίνους, δεν ξέρω αν είναι εδώ, την το ECR. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί, ας είναι λίγο πιο ήπια τα πράγματα από ό,τι ήταν στην αρχή, ελπίζω. Η φιλελευθερωποίηση, η απελευθέρωση είναι αυτό που αποφασίσαμε, όμως ο τίτλος είναι διαφορετικός, είναι η οργάνωση των λιμένων. Υπάρχουν τρία σημεία, τα οποία βέβαια δεν θεσπίζουν κάποια πολύ ιδιαίτερα ε, φοβερά μέτρα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την οδηγία ε, γιατί είναι λίγο πιο ε, πέρα από ότι είχαμε φτάσει για την μεταφορά των υπηρεσιών. Για το θέμα επίσης του δεύτερου κεφαλαίου από όπου βγήκε το θέμα αυτό μετά λόγω των ε, εθνικών προβλημάτων, λόγω των σημαίων. Ε, για τα ρημουλκά και τα λοιπά. Ε, νομίζω ότι αυτό στην ουσία μας έφερε στο να καταρρεύσει η πρόταση και οι Γάλλοι συνάδελφοι επέμεναν ιδιαίτερα. Το θέμα είναι ότι δεν χρειάζεται να έχουμε οπωσδήποτε την εθνική σημαία αφού είναι σε ευρωπαϊκό έδαφος. Πρέπει να τηρούνται απλώς οι προδιαγραφές ε, και για τα εργασιακά και για το ατέλη και τα λοιπά. Και τους Επίσης να πω για την αυτονομία των λιμένων ότι η Ισπανική κυβέρνηση ιδιαίτερα και οι Ισπανοί συνάδελφοι είχαν ένα πρόβλημα γιατί τα τέλη των λιμένων θέλουν σε κάποια ποσοστό να τα ορίζουν από τη Μαδρίτη. Αυτό δεν οδήγησε κατά τη γνώμη μου στο τέλος σε έναν καλό συμβιβασμό, όπως θα έπρεπε τουλάχιστον. Η γαλλική και η ιταλική κυβέρνηση νομίζω λοιπόν με αυτόν τον τρόπο είχαν τη δυνατότητα να παρέμουν και αυτές. Θα πρέπει λοιπόν μετά το καλοκαίρι να ε, εργαστούμε από αυτού του θέματος, ε, να κάνουμε πιο ισορροπημένες αιτιολογικές ε, σκέψεις και μέχρι την ψηφοφορία να μην ψηφίσουμε πριν το δεύτερο, τη δεύτερη ψηφοφορία του DG Competition, γιατί ελπίζουμε η δεύτερη πρόταση να είναι καλύτερη από την πρώτη, αλλιώς θα είναι δύσκολο να ψηφίσουμε. Η Ολλανδή, ε, επίση ε, υπουργό Μεταφορών και ο Επίτροπος για την ανταγωνισμό μου έδωσαν δύο-τρία σημεία τα οποία θα αλλάξουν μάλλον, όμως δεν είναι η Κομισιόν. Ε, δεν είναι αυτή με τους οποίους μιλάμε, αλλά η Κομισιόν. Και πολλές φορές βλέπουμε ότι εμείς κάτι αποφασίζουμε, αλλά τελικά με μονομερή δράση της Κομισιόν αυτά καταστρέφονται. Αυτά. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή και όλους όσοι συνεισέφεραν ώστε να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Με αυτό κλείνει η σημερινή συνεδρίαση και θα συνεχίσουμε και κλεισμένων των θυρών. Να πω κάτι πριν. Έχουν καταρρεύσει και τα δύο πακέτα για τους λιμένες. Ο κύριος ε, Φλέκενστάιν δεν κατέφερε 100% αυτό που ήθελε, αλλά είχαμε καλό συμβιβασμό. Ε, βέβαια αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι εκπροσωπούσε τη θέση του Κοινοβουλίου αλλά ήταν και ικανός να συμβιβαστεί, να έχουμε την διαφάνεια, τα ίδια κριτήρια, τους ίδιους κανόνες αλλά και διαφορετικότητα των λιμένων. Αυτή τη φορά ακούστηκε λοιπόν ο εισηγητής παρόλο που τις άλλες φορές δεν τα κατάφερε. Ευχαριστούμε πολύ για την ε, παρέμβασή σας. Ε, είναι καλό να επενούμε κάποιον. <clears throat> Ευχαριστώ. Ένα σύντομο διάλειμμα και μετά συνεχίζουμε και κλεισμένο τον